Ε, από τον κύριο Ιτουργκάης της... Ε, αναφοράς του, της έκθεσής του για... Ε, ναι. την ετήσια τα πεπραγμένα του 2009 που αφορούν στην Επιτροπή μας. Παρακαλώ τον κύριο Ιτουργκάης να αρχίσει. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ. Όπως ε, είπατε στους συναδέλφους της Επιτροπής, είναι ετήσια έκθεση για τις αποφάσεις της Επιτροπής ε, ε, Αναφορών ε, την προηγούμενη χρονιά και εγώ επίσης είχα το έργο να συντάξω μια έκθεση παρόμοια πριν από αρκετά χρόνια και με υποστήριξε η Γραμματεία. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τη Γραμματεία, την Αλήν και τη βοήθειά της και για μια έκθεση υπάρχει και η μετάφραση την έχετε στα χέρια σας και ταυτόχρονα θα ήθελα να ευχαριστήσω την Έλενα Μάρτιν ε, που βοήθησε στην έκθεση αυτή. Τα σημαντικότερα σημεία σε αυτά που αναφέρομαι φέτος για το 2009 νομίζω ότι χρειάζεται να τονίσουμε ένα γεγονός ότι δεν ήταν ε, μια κανονική χρονιά του Κοινοβουλίου, αλλά κάτι το έκτακτο. Είχαμε τις ευρωεκλογές τότε κάπου εκεί στη μέση και την θέση ισχύ της συνθήκης Λισαβόνας. Η έκθεση του 2009 προσπαθεί να προσφέρει μια σαφή εικόνα των δραστηριοτήτων μας τη χρονιά αυτή και μια εξήγηση πιο συγκεκριμένη τι σημαίνει υποβολή μιας αναφοράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπως επίσης που ενδεχόμενα θα καταλήξει αυτό τις δυνατότητες αλλά και τους περιορισμούς. Ε, εδώ με τη στατιστική ας πούμε για τις διάφορες αναφορές που εξετάσαμε, που μεταβιβάσαμε κλπ. Και, και σε σχέση με τις χώρες και τις υποθέσεις διάφορες. Και υπάρχει μια ποσότητα εργασίας να δούμε και ακριβώς ε, την ε, αξία της εργασίας μας και επίσης τις σχέσεις μας με άλλα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με διάφορα περιφερειακά όργανο και με ανταλλαγές που επηρέασαν τις δραστηριότητές μας. Το 2009 είχαμε κάπως περισσότερες αναφορές από ότι το 2008. Το 2008 είχαμε 1849 αναφορές και το 2009 είχαμε 1924 αναφορές που έφτασαν στα χέρια μας και οι αναφορές ηλεκτρονικά που έφτασαν. Αυτό είναι σημαντικό γεγονός γιατί το 65 περίπου των αναφορών που έφτασαν στα χέρια μας έφτασαν στα χέρια μας ηλεκτρονικά αντί για το 60% του 2008 και επίσης περισσότεροι αναφέροντες που απευθύνονται στο Κοινοβούλιο για θέματα που δεν είναι αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όμως όπως τις συντάξεις, τον υπολογισμό τους και μετά η εφαρμογή δικαστικών αποφάσεων είτε η τον παθητικό χαρακτήρα που δείχνουν διοικητικές υπηρεσίες της χώρας τους ε, και προσπαθούμε, διπλασιάσαμε την προσπάθειά μας για να ενημερώσουμε τους πολίτες για τις αρμοδιότητές μας και θα ήθελα αυτό να το τονίσω στην έκθεση. Το τονίζω λοιπόν. Θα πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες ότι όλα αυτά είναι στα πλαίσια της εφαρμογής των ευρωπαϊκών ρυθμίσεων στα κράτη-μέλη και η Επιτροπή Αναφορών δεν μπορεί να ασχοληθεί με θέματα ε, που υπάρχει μια έρευνα, μια ε, διαδικασία δικαστική, ούτε και να αμφισβητήσει τις δικαστικές ε, αποφάσεις. Εδώ λοιπόν από τη στιγμή που οι εθνικές αρχές έχουν υιοθετήσει μια οριστική απόφαση θα πρέπει όσο γίνεται νωρίτερα ας πούμε σε θέματα περιβάλλοντος να ζητηθεί να εφαρμόσουν οι εθνικές αρχές όλα αυτά που θεωρούνται κατάλληλα ε, στην ρύθμιση την ευρωπαϊκή παραδείγματο χάρη και επίσης ζητάμε να υπάρχει μια περιοδική ενημέρωση για το σε ποιες φάσεις βρίσκονται αυτές ε, οι διαδικασίες επί παραλήψη σχετικά με παρόμοιες υποθέσεις. Ε, να σας πω σε όλους ότι χαιρόμαστε, όπως το είπα στην αρχή, για τη θέση ισχύ της συνθήκης της Σαβώνας ε, και θεωρούμε ότι όλα αυτά θα βοηθήσουν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για πρωτοβουλίες για τους πολίτες και να έχουμε την εγγύηση για περισσότερη διαφάνεια και ευθύνη στη λήψη αποφάσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Ευρωπαίοι πολίτες να μπορούν να υποδείξουν προσθήκες ή αλλαγές στην ίδια την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα λοιπόν με ικανοποίηση δεχόμεθα, υποδεχόμεθα το πράσινη βίβλο της Επιτροπής ε, τέλος του 2009 είναι ένα πρώτο μέρος, πρώτο βήμα εφαρμογής αυτών. Επίσης υποδεχόμαστε θετικά τον δεσμευτικό χαρακτήρα την χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων μετά από τη θέση ισχύ της ε, συνάς και όλα αυτά που χρησιμεύουν για να καταλάβουμε ακριβώς ποια είναι τα θεμέλια δικαιώματα και να τα κατανοήσουν ε, οι πολίτες. Ε, σε προηγούμενη αναφορά για την ε, πραγματοποίηση μιας αναθεώρησης πλήρους των διαδικασιών προσφυγής που έχουν υπόψη τους, που έχουν διάθεσή τους ε, οι πολίτες Ευρωπαϊκής Ένωσης και το πρόσφατο ψήφισμα 9 Φεβρουαρίου του 2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε μια συμφωνία πλαίσιο ανάμεσα στην Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την επόμενη θητεία του Κοινοβουλίου θα εξυπηρετήσει για παρόμοιο σκοπό. Επίσης να σας ενημερώσω για κάτι. Στην έκθεση αυτή εμείς ε, παραπονιόμαστε γιατί δεν ικανοποίησε η Επιτροπή τα δικά μας τα αιτήματα να υπάρχουν επίσημες ενημερώσεις, περιδικές ενημερώσεις για το πώς προχωρούν οι διαδικασίες επί παραλήψη σε σχετικά με ανοιχτές ε, αναφορές που θυμάστε και εμείς οι συντονιστές πολλές φορές ασχοληθήκαμε με αυτές. Επαναλαμβάνουμε λοιπόν ε, ρίσιο ότι είμαστε πεπισμένοι ότι θα πρέπει να απολαμβάνουν διαφάνεια οι πολίτες Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, ακόμα και σε επίσημη διαμαρτυρία όπως επίσης και σε αναφορά σε μας ε, να επαγρυπνεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ώστε να εξετάζονται καλύτερα ακόμα οι αναφορές αυτές και επίσης από τη γραμματεία και από τις πολιτικές ομάδες ζητάμε την επεξεργασία μιας ε, αναθεωρημένης έκδοσης των ρυθμίσεων της εσωτερικής διαδικασίας στην Επιτροπή αναφορών και αυτό θα βοηθήσει και τους βουλευτές στην εργασία τους αλλά θα έχουμε και περισσότερη διαφάνεια στην όλη διαδικασία που ακολουθούμε για τις ε, αναφορές. Να τονίσω ότι θα πρέπει να εργαστούμε και πάνω στη διαφάνεια της διαχείρισης των ίδιων των αναφορών. Εδώ, μέσω της πλήρους πραγματοποίησης και εφαρμοτής ε, αυτό περί αναφορών για μία πρόσβαση των βουλευτών στο αρχείο αναφορών και επίσης ε, ένα site ε, στο ίντερνετ διαδικτυακό ώστε να μπορεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να έχει καλύτερη επαφή με τους πολίτες και να κατανοούν έτσι και τι σημαίνουν ας πούμε ψηφοφορίες και οι υπόλοιπε ενέργειες ε, εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην Επιτροπή μας. Ε, επίσης ε, να δούμε για τις μη αναφόρες. Θεωρούμε ότι θα μπορούσε να υπάρξει μια λύση στην αναθεώρηση της μηχανισμού καταγραφής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και υπεύθυνοι να προσφέρουν τα αρχεία αυτά ε, και μέσω της δική μας Επιτροπής τους πολίτες. Ε, τα μέλη της Επιτροπής αρκετές φορές ε, ρωτήθηκαν για τις μη αναφορές. Πολλές φορές είναι μια άχρηστη απώλεια χρόνου και εδώ θα πρέπει να διαχωρίσουμε εκείνες που κρίνονται απαράδεκτες γιατί είναι στα πλαίσια αρμοδιοτήτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και η Επιτροπή Αναφορών θα πρέπει να προσπαθήσει ακόμα περισσότερο για να εξηγήσει στους πολίτες τι σημαίνει η υποβολή αναφορά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπως επίσης και όλη η διαδικασία καταγραφής αυτών να βελτιωθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και επίση, ολοκληρώνοντα να πω ότι συμμετέχουν ακόμα περισσότερο τώρα τα κράτη-μέλη στις δραστηριότητες της Επιτροπής Αναφορών, όπω επίσης και οι εκπρόσωποι του είναι παρόντε στι συναντήσεις μας. Επίσης τον κεντρικό ρόλο ακριβώς της Επιτροπής και εκτελεστικής και μαζί τους συνεργαζόμαστε για να δούμε αυτές τις παραβιάσεις ενδεχόμενα και να δούμε και αναγνωρίζουμε τις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να μειωθεί ο χρόνος ο συνολικός απάντησης για αιτήματα εξέταση αυτών των θεμάτων που υποβάλλουμε εμείς. Κυρία Πρόεδρε, αυτό είναι κάποιο, κάποιο τρόπο ο απολογισμός, η σύνοψη, η περίληψη προκαταρτικά αυτού του σχεδίου έκθεσης και η γραμματεία αν θέλετε. Ο κ. να μας πει και για την προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών μέχρι πότε θα ισχύει αυτή η προθεσμία και μετά έτσι ανάλογα να δούμε τι θα γίνει και αυτό να πάει μετά στην Ολομέλεια και να ψηφιστεί οριστικά στην Ολομέλεια. Νομίζω ότι θα μπορούσε αυτό αν αληθεύουν οι πληροφορίες μας και οι υπολογισμοί μας ότι πώς να γίνει στην Ολομέλεια του Ιουλίου. Ευχαριστούμε πολύ ε, συνάδελφε. Ε, νομίζω ότι πρέπει να δώσουμε το λόγο τώρα στην Επιτροπή, στην κυρία, στον κύριο Κάσμαν. Ε, παρακαλώ τον κύριο Κάσμαν να λάβει το λόγο. Ευχαριστώ. Thank you, Madam Chair. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ πάρα πολύ και το συνάδελφό σας ε, για μια πολύ ενημερωτική έκθεση και απλώς ως φιλικός παρατηρητής που είμαι εδώ για να βοηθήσω θα αναφερθώ σε δύο από τα τελευταία ζητήματα τα οποία αναφέρατε, συγκεκριμένα τις μη αναφορές και την συμμετοχή των αρχών των κρατών μελών. Εμείς χαιρετίζουμε όλο ιδιαίτερος, ε, όλος ιδιαίτερος την αύξηση της συμμετοχής των ε, αρχών των κρατών μελών και πιστεύουμε ότι είναι ειδικότερα ε, ήταν κυρίως ιδιές, υγιές ε, για τα ζητήματα, για παράδειγμα, περιβάλλοντος και ε, τα κοινωνικά ζητήματα. Όσον αφορά τώρα το θέμα των ε, μη αναφορών, Πιστεύουμε ότι μπορούν πολλά να γίνουν βελτιώνοντας την πρόσβαση. Οι μη αναφορές συνήθως υποβάλλονται ηλεκτρονικά καταλαβαίνουμε το πρόβλημά σας, γιατί και για μας είναι πολύ δύσκολο να τις ε, διαχειριστούμε. Είναι πολύ δύσκολο να διαρθρώσουμε την πρόσβαση των αναφερόντων και αυτό είναι μια πολύ καλή ιδέα. Είναι κάτι το οποίο εμείς κάνουμε, λειτουργεί και είναι κρίμα πραγματικά αν ε, οι αρχές του Κοινοβουλίου δεν διαθέτουν τους απαραίτητους πόρους ε, για να ε, γίνει κάτι τέτοιο. Δεν νομίζω ότι κανένας από τους αναφέροντες που ήταν εδώ εχθές θα είχε αποθαρρυνθεί από μία πιο δύσκολη πρόσβαση για το αίτημά του. Ε, κύριε Όκεν το λόγο. Όκεν. <clears throat> Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Ιτουργκάης για την ε, έκθεσή του, η οποία είναι εξαιρετική. Και θα ήθελα ευθύς αμέσως να περάσω σε ερωτήσεις. Δύο σημεία ήθελα να θέσω. Το πρώτο είναι το case στο οποίο μπορούμε να διαβάσουμε ότι δεν χρειάζεται να ασχολούμαστε με ζητήματα τα οποία, των οποίων μπορούν να επιληφθούν ε, τα ε, δικαστήρια. Εγώ στην ε, εκδοχή του δικού μου κειμένου είναι K. Είναι το K. Είναι το γράμμα K. Στην δική μου εκδοχή του κειμένου βέβαια. Θα συνεχίσω τώρα στα δανεικά. Μπορούμε λοιπόν να διαβάσουμε σε αυτό το σημείο στο οποίο αναφέρθηκα ότι δεν μπορούμε να ασχολούμαστε με ζητήματα με τα οποία ασχολούνται τα εθνικά δικαστήρια. Συμφωνώ, αλλά οι αρμοδιότητες μας ε, είναι κυρίως αρμοδιότητες ε, μεσάζοντο. Ε, δηλαδή μπορούμε να γνωρίζουμε πολύ καλά τι συμβαίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σαφώ βέβαια ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής για παράδειγμα έχει πολύ συγκεκριμένε και περιορισμένε αρμοδιότητε, αλλά υπάρχουν και ορισμένα ε, ζητήματα ε, αστικά, αστικού δικαίου. Και ίσως θα έπρεπε να μπορούσαμε ε, να κάνουμε κάτι ώστε να μην χρειάζεται να φτάνουν τα ζητήματα στη δικαιοσύνη κάθε φορά. Για παράδειγμα, στην Ισπανία πολλές φορές τα δικαστήρια έχουν να αντιμετωπίσουν πληθώρα τέτοιου είδους ζητημάτων και Συνεπώ, πράγματι ισχύει το γεγονό ότι δεν μπορούμε να ασχολούμαστε με όλα αυτά τα ζητήματα. Δεύτερο, πολύ σημαντικό, δεν καταλαβαίνω πολύ καλά γιατί δεν αναφερθήκαμε σε πολύ συγκεκριμένες υποθέσεις ε, με τις οποίες ασχοληθήκαμε, ε, των οποίων ε, επιληφθήκαμε και που δίνουν τη δυνατότητα στον πολίτη να καταλάβει με τι ασχολείται η Επιτροπή μας, ποιες είναι οι εργασίες της και ποιες είναι οι αρμοδιότητές της. Νομίζω ότι είναι πραγματικά πολύ αφηρημένο το να μιλάμε απλώς για τις αρχές θα ήθελα να αναφέρονται συγκεκριμένα παραδείγματα, συγκεκριμένες υποθέσεις. Εγώ μπορώ να σας κάνω έναν ολόκληρο κατάλογο αν θέλετε. Νομίζω ότι χρειάζεται ένας κατάλογος που να δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες να καταλαβαίνουν γιατί πράγμα μιλάμε. Πρέπει να μπορούμε να στραφούμε προς τους πολίτες και να τους πούμε να αυτά έχουμε καταφέρει να κάνουμε. Πρέπει να είμαστε πιο φιλικοί προς τον πολίτη για να το πω έτσι. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και εγώ κυρία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 Ευχαριστώ πολύ και εγώ θα ήθελα να πω ότι είναι μια εξαιρετική έκθεση για μια πολύ δύσκολη περίοδο μετάβαση από τη μία κοινοβουλευτική θητεία στην άλλη και υπήρξαν και πολλές ε, αλλαγές ε, στο πλαίσιο της δικής μας Επιτροπής. Ε, οι συνεργασίε μας όμως συνεχίστηκαν με πολύ ομαλό τρόπο. Επίσης έχουμε και μία νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή και γνωρίζουμε ότι ο ρόλο Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι πολύ σημαντικός για τη δουλειά μα. Οπότε, ευχαριστούμε πολύ για για την έκθεση και ευχαριστούμε πολύ για ε, την ομαλή ε, έκβασή της. Θα ήθελα να τονίσω περαιτέρω κάτι το οποίο αναφέρετε κι εσείς. Για παράδειγμα, το αίτημα των, της διαφανούς λειτουργίας και με πιο προσανατολισμένης προς τον πολίτη λειτουργία των ευρωπαϊκών οργάνων. Αυτό το ζήτημα του προσανατολισμού προς τον ε, πολίτη, άμα το τονίζαμε περισσότερο, θα ήταν πολύ χρήσιμο. Επίσης, την ανάγκη βοήθειας από τους ε, επιτρόπους ε, και αυτό θα ήταν πολύ χρήσιμο. Κάτι ακόμη θα ήθελα να τονίσω, μεταξύ αυτών που αναφέρεται, την έναρξη των διαπραγματεύσεων για μια νέα διοργάνωση Ιρανική Συμφωνία θα είναι απολύτω απαραίτητη λόγω τη αυξημένη ε, σημασία των δικαιωμάτων των πολιτών. Το αναφέρετε και εσεί στη Χάρτα των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, στο πλαίσιο τη Συνθήκη Λισαβόνα κλπ. Και, επίση και θα είναι πολύ σημαντικό να ε, επεξεργαστούμε έναν αναθεωρημένο οδηγό για ε, τα μέλη της Επιτροπής μας, ε, του εσωτερικού κανονισμού, για να γνωρίζουν ακριβώς τα μέλη της, τον κανονισμό. Επίσης είναι πολύ ενδιαφέρον το γεγονός ότι πολλές χώρες, ότι από πολλές χώρες όπως για παράδειγμα Γερμανία, Ρουμανία, Ιταλία, προέρχονται πολλές αναφορές. Είναι ένα θετικό μεν μήνυμα, αλλά υπάρχει και και αρνητικό μήνυμα που θα μπορούσαμε να λάβουμε από αυτό. Γιατί δεν λαμβάνουμε περισσότερε αναφορέ από άλλε χώρε. Μπορεί να σημαίνει ότι υπάρχουν λιγότερα προβλήματα, αλλά μπορεί να σημαίνει ότι υπάρχει και χαμηλότερο επίπεδο γνώσης ε, των δικαιωμάτων του πολίτη. Και ίσως θα έπρεπε να επικεντρωθούμε περισσότερο στις χώρες αυτές ε, από τις οποίες λαμβάνουμε λιγότερες αναφορές. Θα μπορούσαμε να διερευνήσουμε περισσότερο το ζήτημα ε, των λόγων για τους οποίους συμβαίνει αυτό. Επίσης συμφωνώ απολύτως με τη δήλωσή σας που είπατε ότι η επίσπευση της απάντησης ε, της Επιτροπής μας ε, ε, είναι χρήσιμη γιατί καμιά φορά όταν αργεί η απάντηση μπορεί να απογοητεύονται και να αποθαρρύνονται οι πολίτες όπως για παράδειγμα με τις διαδικασίες επί παραβάση που πολλές φορές είναι πολύ αργές και δεν αποτελούν πραγματική κατάλληλη απάντηση προς τους, πολιτέ, πολίτες. Και δεν, δεν ξέρω μήπως θα μπορούσαμε να βελτιώσουμε ολόκληρη τη διαδικασία. Όσον αφορά τώρα τα παράπονα των πολιτών ε, και την ε, ανάπτυξη της, της ιστοσελίδας ε, EU Rights, δικαιώματα στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι κάτι το οποίο θα μπορούσε να βοηθήσει πολύ για να λαμβάνουμε τις αναφορές με καλύτερο τρόπο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Γκέντς. Κυρία Wallis. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε και ευχαριστώ πολύ τον εισηγητή, τον κύριο Ιτουρκάης ε, για ε, την ε, πολύ καλή και περιεκτική του έκθεση. Θα ήθελα να επικεντρωθώ σε δύο ζητήματα. Ήδη πολλά υπόθηκαν για το κατά πόσο η προσέγγιση μας πρέπει να είναι φιλική προς τον πολίτη. Είναι ένα ζήτημα συνεχώς ε, τα, τα τελευταία έτη και θέλουμε πάντοτε να το προωθήσουμε, να υπάρχει μεγαλύτερη συνοχή στον τρόπο με τον οποίο μας προσεγγίζουν οι πολίτες, να γνωρίζουν πού ακριβώς πρέπει να, έρθουν. Ε, η ενιαία θηρίδα, εν πάση περιπτώσει, αντί, να, ε, αντί να πρέπει ο πολίτης να πάει είτε σε εμά είτε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το ζήτημα είναι τώρα η αναδιάρθρωση αυτό που κι εσείς αναφέρετε, ε, η μονάδα ε, αλληλογραφίας των πολιτών είναι κάτι το πάρα πολύ ε, χρήσιμο γιατί θα βελτιώσει την πρόσβαση των πολιτών σε εμά. Κάτι ακόμη, ακούγοντας την παρουσίασή σας και ακούγοντας τα σχόλιά σας μετά την έναρξη ισχύω της συνθήκης της Λισαβόνας, Υπάρχει κάτι που θα μπορούσαμε να κάνουμε περισσότερο. Κατά τη διάρκεια των συζητήσεων μεταξύ των ε, οργάνων για την νέα ε, συμφωνία πλαίσιο υπήρχε συζήτηση ε, υπάρχει Υπάρχει αναφορά κυρίως στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γνωρίζουμε όμως ότι ε, οι επαφές μας με τα κράτη-μέλη είναι ακόμη σημαντικότερες για την επίλυση ορισμένων προβλημάτων. Υπάρχει όμως και ένας άλλος τρόπος προσέγγισης του ζητήματος αυτού και επομένως ε, ο τρόπος είναι πολύ πιο στενή σχέση ε, σε επίπεδο κοινοβουλίου. Υπάρχουν πολλές επιτροπές αναφορών και σε εθνικά και σε περιφερειακά κοινοβούλια και νομίζω ότι θα έπρεπε να συνενώσουμε τις δυνάμεις μας και τον αγώνα μας μαζί τους γιατί αυτό θα αντιμετωπίσει το ζήτημα των μη αναφορών. Αν ε, φτάνουν δηλαδή σε λάθος επίπεδο διακυβέρνηση για να το πω έτσι. Θα ήθελα λοιπόν να συμπεριληφθεί κάτι που θα αναφέρει ε, αυτόν, αυτήν την κατεύθυνση. Έχουμε κάνει προσπάθειες ε, στο παρελθόν, αλλά μετά τη Λισαβόνα υπάρχει πολύ καλύτερη βάση και δομή για να το κάνουμε αυτό και ενδεχομένως να απαντήσει εν μέρη στο ερώτημα ε, των χωρών από τις οποίες δεν λαμβάνουμε πολλές ε, αναφορές. Μπορεί να μην έχουν ε, πολλές, πολύ δραστήριες επιτροπές αναφορών. Είναι κάτι το οποίο θα έπρεπε περισσότερο να διευνήσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Βέβαια θα πρέπει να απαντήσουμε γιατί από το Λουξεμβούργο έχουμε τόσο λίγες αναφορές. Είναι επειδή δεν είναι ενημερωμένοι ή επειδή δεν έχουν προβλήματα. Αυτό είναι ένα τέτοιο είναι ένα ζήτημα που θα πρέπει να ερευνηθεί. Η κυρία, ο κύριος Μέιερ παρακαλώ. Ε, Ευχαριστώ πρόεδρε. Να ευχαριστήσω τον κύριο Ιτουργκάης γιατί η έκθεση αυτή είναι πλήρης, ιδιαίτερα πλήρης και λεπτομεριακή. Να τονίσω επίσης ορισμένες πτυχές εκεί που έχει σημασία αυτό για τις απαντήσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής για διάφορες υποθέσεις που μας κάνουν και καθυστερούμε αυτές οι καθυστερήσεις και εμείς με τη σειρά μας ε, θα ήθελα να σας πω ότι όταν θέλουμε να έχουμε στα οικοσυστήματα ευρωπαϊκά άμεσες ε, αρμοδιότητες και, στην, ε, και για το περιβάλλον αυτό τις αρμοδιότητες μας ε, τι κάνουμε για αρμοδιότητες για την εφαρμογή για την προστασία των υδάτων, του περιβάλλοντος κλπ. Τα τελευταία πέντε χρόνια τι έγινε. Οι διάφορες διαδικασίες επί παραλήψη πολλές φορές ξεκινάνε αργά δηλαδή πραγματοποιείται ένα έργο δημόσιο ιδιωτικό σε κάποιο κράτος μέλος και δεν σέβεται διάφορες οδηγίες ευρωπαϊκές να που συντάσσεται η αναφορά φτάνει εδώ, μας λέει την απόψη της Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τώρα μέχρι να γίνουν όλα αυτά πράγματα, μέχρι να φτάσει από εδώ από εκεί, να πάει στο κράτος μέλος ε, και ότι δεν σέβονται κλπ περνάει τόσος χρόνος που μέχρι τότε έχει τελειώσει το έργο. Άρα λοιπόν ε, δεν μπορούν να διορθωθούν πια οι ζημιές. Γι' αυτό κύριε Τουργκάης, να πούμε ότι θα πρέπει να το τονίσουμε αυτό που ήδη το αναφέρετε εσείς στην έκθεσή σας, ότι θα πρέπει η διαδικασία να είναι πιο σύντομη, κυρίως όταν πρόκειται για δημόσια ή ιδιωτικά έργα που επειδή είναι σημαντικά μπορούν να βλάψουν ιδιαίτερα το οικοσύστημα. Έτσι, γιατί αν καθυστερούμε, έστω και αν έχουμε τις αρμοδιότητες, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα στο κάτω, στο τέλος τέλος για να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Ε, θα πρέπει το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο κλπ. να προστατεύουν και να ερευνούν για την τήρηση των ρυθμίσεων των ευρωπαϊκών. Πολλές φορές όλα αυτά φτάνουν αργά, δικαστικές αποφάσεις που καθυστερούν και όταν εκδοθεί απόφαση έχει γίνει πια η ζημιά και ακόμα και αν υπάρξει μια οικονομική αποζημίωση δεν διορθώνει τη ζημιά. Για τον κύριο Τουργκάης λοιπόν θα μπορούσε να συμπληρώσει έτσι το μέρος αυτό που αναφέρθηκε από το μέρος και ασκή κριτική και να ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, μεγαλύτερη για ταχύτητα στην απάντηση αυτό για να μπορέσουμε να αποφεύγουμε παρόμοιες ζήμιες. Αυτό Ολοκληρώντα να ευχαριστήσω τον κύριο Τουργκάης που συνέταξε μια καλή νομίζω έκθεση και έχει μια συνολική, δίνει μια συνολική εικόνα, μια προς μια άποψη των όσων έχουν γίνει και των βελτιώσεων όπως επίσης και το site το ηλεκτρονικό ακριβώς που λέει και ο Σιτουργκάης θα πρέπει να ενισχυθεί γίνουν και περισσότερο οι Ευρωπαίοι πολίτες ηλεκτρονικά απευθύνουν σε εμά την αναφορά τους άρα λοιπόν να βελτιώσουμε το τρόπο αυτό μεταβίβασης και έτσι με τη συμμετοχή περισσότερο του πολίτου. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μέγερη. Κύριε Μινάς, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε να ευχαριστήσω τον κύριο Τουργκάης για την έκθεση του και όπως είπε ο Βίλι Μέγερ για να μπορέσουμε να τη συμπληρώσουμε αυτή την έκθεση, να είναι καλύτερη επικεντρωμένη, αντικειμενική, θα πρέπει να δούμε στο διατακτικό ακριβώς ορισμένα πράγματα που δεν έχουν γίνει με εκθέσεις ή που έχουν κλείσει χωρίς να γίνει κάτι. Να εξηγήσουμε ότι έχουμε τόσες αναφορές, αλλά από αυτές τις αναφορές μέχρι και το 46% από ό,τι λέγεται στο στο εισαγωγικό δεν κρίθηκαν παραδεκτές. Και λοιπόν θα πρέπει να καταλάβει κανείς πως έχει αυτή η κατάσταση στην Ευρώπη, να λέμε ποιες είναι συγκεκριμένε αναφορές ανάλογα με χώρες, με θέματα κλπ. Και αυτά στη αιτιολογική σκέψη και στο κύριο μέρος να δούμε σε τι ακριβώς αναφέρονται αυτές που δεν έχουν γίνει δεκτές προς εξέταση ή που δεν μπόρεσε να εξετάσει το Ευρωκοινοβούλιο η Επιτροπή μας γιατί λέει ότι τόσες ε, ε, απερίφθησαν αλλά δεν αναφέρεται σε ποιες χώρες είναι αυτές ε, από τη Γερμανία πάρα πολλές αναφορές αλλά δεν σημαίνει ότι ο αριθμός τους ε, σημαίνει ότι δεν έχουν να κάνουν με μη Είναι απλά και μόνο αναφορές έτσι γενικά. Άρα λοιπόν όλα αυτά θα πρέπει να αναφέρονται με περισσότερες λεπτομέρειες στην όλη έκθεση του κ. Τουργκάης. Ε, βέβαια αυτό θα έμοιαζε κάτι σαν ε, έρευνα, ε, μια μελέτη ειδική που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί αργότερα από εμάς ε, δεν ξέρω αν σε μια ετήσια αναφορά θα έπρεπε να μπει κανεί σε τέτοιε λεπτομέρειε, αλλά αυτό είναι κάτι που πρέπει ίσω να το συζητήσουμε. Ε, ο Ναι, σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον εισηγητή για την άριστη έκθεσή του. Όλα αυτά χρειάζονται άλλωστε για να δείξουμε ποια είναι η φύση της εργασίας μας. Και όσα είπε η προηγούμενη ομιλήτρια, να πω και εγώ ότι χρειάζεται να αναφέρουμε συγκεκριμένα παραδείγματα, κάτι που μπορεί να ενθαρρύνει τους πολίτες μας, γνωρίζοντας πως έχει κατάσταση, να συντάσσουν τις εκθέσεις τους και να τις απευθύνουν σε μας. Ορισμένα παραδείγματα, ας πούμε, θα εμπλούτιζαν την όλη έκθεση. Και ακόμα σχετικά με όσα είπε ο κ. Μέγερ για το μέρος αυτό το σημαντικό με την άρχιση κάποιες κριτικής κλπ. Εδώ αναφέρεται το πόσος χρόνος περνάει. Εδώ για, για τις μη αναφορές με αφορά προσωπικά το θέμα γιατί αν μπορούσαμε να ξεχωρίσουμε αποτελεσματικότερα και γοργά τις μη αναφορές από τις αναφορές θα μπορούσαμε και καλύτερα να εργαστούμε. Σίγουρα είναι σημαντικότατο το ίντερνετ. Μου αρέσει, με ενδιαφέρει. Αλλά πρέπει βέβαια και οι πολίτες να το χρησιμοποιούν, αλλά αυτό δεν μας βοηθάει και πολύ. Γιατί εντάξει μπορούν όλα αυτά να γίνουν στα γρήγορα, αλλά τι θα γίνει αν δεν μπορέσει να εξεταστεί η σχετική έκθεση. Πρέπει να βρεθεί ένας κάποιος τρόπος για να ξεχωρίσουμε τις ε- αναφορές από τις μη αναφορές και θα πρέπει να δούμε πώς θα μπορούσαμε να έχουμε ταχύτερα απάντηση για εκείνες που εξετάζουμε θα μπορούσαμε ίσως να συντάξουμε ένα κατάλογο με, κατεπήγοντες, με κατεπήγουσες αναφορές και να τις ξεχωρίσουμε από τις υπόλοιπες, εκεί που απαιτείται δηλαδή άμεση γοργή εξέταση. Υπάρχουν περιπτώσεις ας πούμε και ατόμων που γράφουν, ξαναγράφουν, επιμένουν, επαναλαμβάνουν, επανασεντάσουν. και θα ήθελα να πω ότι η... θα πρέπει να συγχαρούμε και μερικές φορές την Επιτροπή και Ευρωπαϊκή αλλά και να τη να είναι και πιο γρήγορες απαντήσεις της. Από άλλη μεριά έχουμε και επίσης και τα κράτη-μέλη που απαντούν με καθυστέρηση. Έχουμε και θετικά παραδείγματα που μπορούμε να συμπεριλάβουμε. Κανονικά θα πρέπει να υπάρχει μια μέθοδος για να ξεχωρίσουμε, να διαχωρίσουμε την αναφορά από τη μία αναφορά και ακόμα κάτι, όπως είπαμε, όσο γίνεται ταχύτερα απάντηση. Ε, εγώ ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε κύριε Γιά. Ο κύριος Κάσπαν θα ήθελε ίσως να ε, απαντήσει σε ε, διατυπώσεις που έγιναν στη διάρκεια από τους συναδέλφους. Thank you, Mr. Ε, ε- Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε για την έκθεση αυτή. Νομίζω ότι μας ε, δίνει σημαντικές πληροφορίες για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει και η Επιτροπή Αναφορών αλλά και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η έκθεση αναγνωρίζει το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι φυσικός εταίρος της Επιτροπής Αναφορών και αυτό αντικατοπτρίζει όχι μόνο το γεγονός ότι προσπαθούμε να ανταποκριθούμε ε, στις ε, ανησυχίες που μας ζητάτε να εξετάσουμε, αλλά και εμείς ε, πρέπει να επιληφθούμε ζητημάτων ε, τα οποία ομοιάζουν ε, με τα θέματα που εξετάζονται στην Επιτροπή Αναφορών. Υπάρχει λοιπόν η ανάγκη να εξηγήσουμε στους πολίτες ε, τα όρια των αρμοδιοτήτων μας, τα όρια των ε, αρμοδιοτήτων της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και τα όρια των εθνικών αρμοδιοτήτων και αυτό για μας συνιστά μια συνεχή πρόκληση. Επίσης, η αναφορά στο περιβάλλον, που είναι κάτι που πολλές φορές απασχολεί τους πολίτες. Ο κύριος Μέγερ αναφέρθηκε στην επίσπευση της, ε, της παρέμβασης. Είναι κάτι βέβαια το οποίο ανησυχεί και εμάς, μας απασχολεί και όσον αφορά τις ε, δυνατότητες ε, που έχουμε εμείς στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι οι προσωρινά μέτρα που μπορούμε να ζητήσουμε από το δικαστήριο σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Για παράδειγμα, Κατά την τελευταία κοινοβουλευτική θητεία πολλές φορές ε, είχαμε τέτοιου είδους προσωρινά μέτρα από το δικαστήριο και το καλύτερο παράδειγμα είναι ενδεχομένω ε, την κοιλάδα Ρασπούτη που ήταν ε, αντικείμενο μίας αναφοράς εδώ στην Επιτροπή σας. Υπάρχουν ιδιαίτερες δυσκολίες και προκλήσεις όταν αναζητούμε προσωρινά μέτρα και νομίζω ότι θα έπρεπε να διερευνήσουμε και άλλες διόδους για να εξασφαλίσουμε ότι αποκαθίστανται τα προβλήματα των πολιτών και γι' αυτό ακριβώς χαιρετίζουμε ιδιαίτερα την αναφορά στο ρόλο των εθνικών δικαστών στο πλαίσιο της έκθεσης αυτής. Εμείς προωθούμε την συνεργασία με τους εθνικούς δικαστές ε, με σκοπό την προώθηση της ε, ευαισθητοποίησής τους ε, για την ευρωπαϊκή νομοθεσία και τη γνώση αυτής. Επίσης βλέπουμε το βαθμό στο οποίο, στο πλαίσιο ενός εθνικού συστήματος, ε, να, μπορεί κανείς να αναζητήσει κάποιο είδους ανακούφιση. Δεν είναι κάτι μόνο ε, που μπορεί να συμβεί μόνο στην, ε, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, μπορεί να συμβεί και σε εθνικό επίπεδο και μερικές φορές αυτό το επίπεδο δικαιολογείται κιόλα. Συχνά κινούμεθα προς την ίδια κατεύθυνση Έχουμε τους ίδιους στόχους ε, να επισπεύσουμε την αποκατάσταση των προβλημάτων το συντομότερο δυνατόν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, να πω κάτι μισό λεπτό. Πάντως ούτως ή άλλως εκτιμώ κύριε Τουργκάης ότι μέσα από την αναφορά σας και όσα υπόθηκαν ε, αυτό που προκύπτει είναι ότι πέρα από την ενεργοποίηση των ε, πολιτών ε, πρέπει να ενεργοποιήσουμε και την Κομισιόν και βεβαίως και τα εθνικά κράτη. Είναι ίσως από τη δράση της Επιτροπής μας θα προκύψουν τέτοιου είδους ε, ε, αποτελέσματα και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. μπορείτε να έχετε το λόγο. Κυρία Πρόεδρε, σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους πήραν το λόγο, όπως επίσης και για τα σχόλιά τους και από την Επιτροπή για αυτές τις μη αναφορές και πώς θα βελτιωθεί το ιστοσελίδα με τον κύριο και τον κύριο Χαρ Για αυτά τα σχόλια τους ευχαριστώ. Ναι. Έχει καταβληθεί προσπάθεια και καταβάλλεται προσπάθεια. Χρειάζεται να συμπληρωθούν αυτές τις προσπάθειες κυρία Επιτροπή είπε ότι κρίμα που δεν προσφέρουν πόρους ε, τα θεσμικά όργανα γι' αυτό. Έτσι, εμείς ε, θα πρέπει να καταβάλουμε κάθε προσπάθεια και μήπως και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να μας βοηθήσει λοιπόν ε, για να βελτιωθούν αυτοί οι τρόποι και να καταλάβουμε ότι μια ιστοσελίδα έχει μεγάλη σημασία και αν ενισχυθούμε, αν ενισχυθεί αυτό θα έχει σημαντικό ρόλο να παίξει και νομίζουμε ότι έτσι τα σχόλια αυτά, όλα αυτά τα επιχειρήματα μπορούν να σταθούν ακόμα περισσότερο με μια, μια επιτυχημένη ιστοσελίδα και βοηθάει την καλή λειτουργία μας αυτή η ιστοσελίδα. Μάργαρετ, ε, συμπίπτει η άποψή της με την Μαρία Μονιθ ότι για περιπτώσεις ε, με συγκεκριμένες υποθέσεις ε, που θα πρέπει να ληφθούν υπόψει και όχι αφηρημένα πράγματα. Γιατί δεν ανέφερα κάτι συγκεκριμένο στις διάφορες προηγούμενες εκθέσεις κάθε χρονιά δεν μπήκαμε σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, δεν αναφέραμε συγκεκριμένες αναφορές. Αλλά εντάξει, όπως καταλαβαίνετε, Είμαι στη διάθεσή σας και μπορώ να το αλλάξω αυτό. Μπορούμε να φέρουμε συγκεκριμένα παραδείγματα, εάν πιστεύετε βέβαια ότι κάτι τέτοιο θα ήταν καλύτερο και για τους ίδιους τους αναφέροντες. Ε, και να υπάρχει ένας κάποιος οδηγός για να σε εισαγωγικά να περπατούν καλύτερα για να κάνουν αυτό που θέλουν να συντάξουν ε, και έτσι να αλλάξουν τα πράγματα για να υπάρχει ένα συνδυασμό διαφόρων συναφών περιπτώσεων και να μπορέσει ε, να, να, σε αυτές τις περιπτώσεις ε, όπως είπαμε. Η κύριε Μπονς μίλησε για τη δύσκολη περίοδο εδώ στην Επιτροπή λόγω των αλλαγών των μεταβολών εδώ στην Επιτροπή Μεταφορών θα τα θυμάστε όπως η κυρία Γκόνς, ας πούμε, καταλαβαίνει ότι έχει μεγάλη σημασία εδώ η Επιτροπή και προς αυτήν την κατεύθυνση πηγαίνουν τα σχόλιά της. Επίσης ένα σχόλιο ιδιαίτερα ενδεικτικό που είπε ότι θα πρέπει οι επίτροποι να τα καταλάβουν αυτά, οι καινούργοι τουλάχιστον. Ε, δεν ξέρω τι γίνεται όμως όταν υπάρχει μια υπογραφή ε, κάποιου άσχετου δεν μπορούμε να είμαστε εμείς άσχετοι που θα ασχοληθούμε αυτά. Έχουμε σημασία, έχουμε ένα ρόλο να παίξουμε και εδώ οι πρωταγωνιστές επίσης είναι οι πολίτες της Ευρώπης και αλλού σε περιφερειακά κοινοβούλια, αστυνομικά κοινοβούλια δεν μπορούν να πάνε και Εδώ μπορούν να έρθουν και να εξιστορήσουν τα προβλήματά τους, να συζητήσουν με την Επιτροπή, με τους Ευρωβουλευτές και θα πρέπει και οι ίδιοι η Επιτροπή και οι πολιτικοί να καταβάλουν μια προσπάθεια να διευκολύνουν τη δυνατότητα αυτή των Ευρωπαίων πολιτών για να μας γνωστοποιήσουν τα προβλήματά τους οι πολίτες ακριβώς. Επίσης, γιατί από ορισμένε χώρες δεν έχουμε περισσότερες αναφόρες και περισσότερες φορές είναι η Ισπανία, το με η Ιταλία, Ιταλία, Γερμανία, από εκεί είναι οι πολλές αναφόρες. Ίσως όμως αυτό συμβαίνει επειδή εκεί υπάρχουν 90 εκατομμύρια ε, κάτοικοι στο μία χώρα και απ' την άλλη δεν έχουμε ούτε ένα εκατομμύριο. Ίσως παίζει και αυτό ρόλο λοιπόν. Και επίσης ε, για τα σχόλια, για τα ποσοστιαία για τα εκατοστία ποσοστά. Εντάξει, δεν τα ανέφερα αυτά γιατί δεν συμπίπτουν τα ποσοστά από τη μία χώρα στην άλλη. Κυρία Βόλης, άκουσα σήμερα, αλλά είχε κάνει ένα σχόλιο, θα ήθελα να το επαναδιατυπώσω εδώ. Είναι σημαντικό να δούμε τις στενές σχέσεις με τα περιφερειακά και εθνικά κοινοβούλια, εκεί που υπάρχουν ήδη επιτροπές αναφορών. Το έχουμε κάνει, δεν ξέρω αν ε, κάποιοι συναδελφοί από την προηγούμενη θητεία, το θυμάται, είχαμε πάει στη Γερμανία, στη Σκοτία, Ζωντεύει, το θυμάται. Λοιπόν, και για τη γραμματεία επίσης, μήπως σε μια κάποια επόμενη συνάντηση, εάν νομίζετε ότι είναι πρέπον, να έχουμε μια... να δούμε με ε, κοινοβούλια, με περιφερειακά κοινοβούλια να μπορέσουμε να καταστήσουμε μια σχέση, να συνεργαστούμε, να ανταλλάξουμε απόψεις σε μια συνάντηση, τι μπορεί να γίνει με αυτές τις επιτροπές αναφορών, τι γίνεται, πώς θα μπορούσε κανείς να έχει μια επαφή και να υπάρχει αυτή η σχέση γιατί δεν έχουμε παντού σε όλες τις χώρες επιτροπή αναφορών υπάρχει κάτι το αντίστοιχο αλλά δεν είναι ακριβώς όπως μια επιτροπή αναφορών Άρα λοιπόν, εντάξει πολλά να θέτουμε στη γραμματεία, αλλά μήπως η γραμματεία θα μπορούσε να ρίξει μια ματιά, καλό θα ήταν διαφωτιστικό για να μπορέσουμε να εργαστούμε. Αν λοιπόν το θεωρεί πρέπει η γραμματεία και το Προεδρείο, yeah. τον φίλο Μέγερ για το χρόνο απάντηση ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ε, παρόλο που η δικαιολογία μας δεν συμπίπτει, αρκετέ φορέ καταφέραμε να πετύχουμε κάτι καλό με τα σχόλιά μας, θα μπορούσαμε να είμαστε συμπληρωματικοί και με το Μέγερ, με το Βιλί θα μπορούσαμε να έχουμε κάτι συμπληρωματικό για το κείμενο αυτό, για την έκθεση αυτή και θα μπορούσαμε έτσι να ακουστεί περισσότερο το κάθε παράπονο που γινόταν για την πολύ καθυστερημένη απάντηση που προσφέρεται και επίσης για την ιστοσελίδα, όλα αυτά που είμαστε στην αρχή, με μια ειδική αντιμετώπιση. Η Μαρία ε, ε, Γιατί το θέμα Μαρία Μουνιά, ε, το είχα πει πιο πριν ότι σε σχέση με τη σύνταξη άλλων εκθέσεων. Αν είναι η πλειοψηφία αυτή δεν έχω κανένα πρόβλημα να το δεχτούμε. Και σε σχέση ευχαριστώ με τα σχόλια τα οποία έγιναν. Και αυτό θα μας βοηθήσει, θα υποστηρίξει τους συντάκτες αναφορών, ώστε να κατανοήσουν πολλές φορές ε, τι συμβαίνει με τις αναφορές που πρέπει να εξεταστούν εδώ, που πρέπει να συνάδουν με το κοινοτικό δίκτυο, δίκαιο, που πολλές φορές δεν ευθυγραμμίζονται με αυτό. Ο κύριος Χάρ στην ίδια γραμμή σχολίασε κάτι και το ίδιο έχουμε ε, κάνει και ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε επίσης τα σχόλια της κυρίας Παλιαδέλη για την λειτουργία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, αν γίνεται τα κράτη-μέλη να, να μπορέσουν να ευθυγραμμιστούν, να μπορέσουμε σε αυτό το σημείο στην Επιτροπή Αναφορών να προαγάγουμε το θέμα. Και πρέπει να πούμε σε σχέση με το θέμα αυτό, να τονίσουμε το ρόλο που διαδραματίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε σχέση με την Επιτροπή Αναφορών. Και αυτά. Ξέχασα ίσως πιο πριν και ίσως ε, αν συμφωνείτε Πρόεδρε να σχολιαστεί το θέμα των τροπολογιών. Ποιες είναι οι προθεσμίες Α, εντάξει, ε, πρωτού ε, αναφερθεί αυτό, μπορείτε εσείς να το κάνετε. Ευχαριστώ. Ευχαριστήσω για την παρουσίαση. Ε, να σας συγχαρώ για την ε, εισήγηση, ε, να σας παρακαλέσω να, έρθει στη θέση μου προκειμένου να προχωρήσει του κ. Μποστινάρου η παρουσίαση της δικής του έκθεσης, γιατί εγώ πρέπει να φύγω, και να κλείσω λέγοντας ότι οι ημερομηνίε για τις τροπολογίες είναι η 6η Μαΐου στις 12 το μεσημέρι. Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί την 1η Ιουνίου στις 10 το πρωί και ε, στην Ολομέλεια ε, του Ιουλίου θα έχουμε την τελική ψήφο από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ε, καλή σας μέρα, εγώ πρέπει να φύγω. Κύριε Κουργκάης, παρακαλώ να προεδρεύσετε του, συνέχεια. Δεν έχω πρόβλημα εγώ, αλλά είναι ο δεύτερος αντιπρόεδρος και εκείνο θα αναλάβει τώρα την προεδρία, παρακαλώ. Okay. Ε, εντάξει, μπορούμε να ξεκινήσουμε τώρα. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Ο κύριο Ιτούργαϊθ να αναλαβανε την Προεδρία. Εν πάση περιπτώσει ομω ακολουθωντα την ημερήσια διάταξη, θα δώσουμε τον λόγο στον κύριο Μποστινάρο σε σχέση με την βιοπικιλότητα ω θέμα που είχαμε την ευκαιρία να έχουμε με πρώτη παρουσία. Σας δίνω τον λόγο κύριε Μποστινάρο. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ξεκινήσω την πολύ σύντομη παρουσίαση συμπερασμάτων με την παρουσίασή μου με τα συμπεράσματα που έχουν συνταχθεί και διανεμηθεί. Απέτυχε η Ευρωπαϊκή Ένωση στο πρώτο πρόγραμμα δράσης της όσον αφορά τη βιοπικιλότητα. Και έτσι αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να συνεχίσουμε τώρα ξεκινώντας μελλοντικές δράσεις ως Ευρωβουλευτές και ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρέπει να επιλύσουμε πρώτα αυτό το πρόβλημα λοιπόν. Η δική μου γνωμοδότηση βασίζεται σε τρία ουσιοδέστερα στοιχεία. Πρώτα απ' όλα χρειαζόμαστε διασυνοριακή συνεργασία. Αυτό είναι το πρώτο. Σήμερα είναι προφανές πρόδειλο ότι χωρίς αυτή τη διασυνοριακή συνεργασία και χωρίς διεθνή συνεργασία δεν θα καταφέρουμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα της ε, καταστροφής, της αποψήλωσης ε, της ε, βιοπικιλότητας. Να σας υπενθυμίσω ότι όταν συζητούσαμε αυτά τα θέματα κάναμε λόγο για δύο μείζωνα θέματα υποδομής το North Stream στην Βαλτική θάλασσα και το South Stream, άλλον αγωγό δηλαδή, στη Μαύρη θάλασσα. Και τώρα ο αγωγός Ναμπούκο έχει εγγραφεί στον πίνακα αναμονής για το 2011. Και αυτά τα τρία προγράμματα ή σχέδια ε, αφορούν κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν εταιρικέ σχέσεις με μη κράτη-μέλη και σε, αυτή την, σε αυτό το πλαίσιο έχουμε και κράτη τα οποία δεν είναι έχουν, δεν έχουν προοπτική, δεν θέλουν να ενταχθούν, δεν πρόκειται να ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά τα εγχειρήματα θα έχουν μεγάλε ε, τεράστιες επιπτώσει στην βιοπικιλότητα. Γι' αυτό χρειαζόμαστε την διασυνοριακή συνεργασία. Οι κανονισμοί και οι προδιαγραφέ, λοιπόν για την προστασία του περιβάλλοντο και για την προστασία τη βιοπικιλότητα πρέπει να είναι υποχρεωτικού χαρακτήρα, δεσμευτικού και υποχρεωτικού χαρακτήρα που θα δεσμεύουν την Ευρωπαϊκή Ένωση και του εταίρους τη. Ε, Δεύτερο σημείο. Χρειαζόμαστε οπωσδήποτε έναν σαφή ορισμό για τις περιόδους ε, ή προθεσμίες αντίδρασης και ανταπόκρισης από τα κράτη-μέλη. Αντίδραση και ανταπόκριση όταν υπάρχει μια αρνητική επίπτωση στην βιοπικιλότητα και χρειαζόμαστε ένα σαφές χρονοπλαίσιο για να μπορέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δραστηριοποιηθεί. Πάντα υπάρχει μια καθυστέρηση όταν αντιμετωπίζουν τέτοιου είδου προβλήματα τα κράτη-μέλη. Υπάρχει καθυστέρηση και στην δράση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και όλες αυτές σορευτικά οι καθυστερήσεις οδηγούν σε ανεπανόρθωτες καταστροφές της βιοπικιλότητας. Μετά υπάρχει ένα τρίτο ουσιοδέστερο σημείο. Το στοιχείο αυτό είναι ότι χρειάζονται αυστηρότερα κριτήρια οπωσδήποτε κριτήρια αυστηρότερα τα οποία θα καθορίζουν την ποιότητα, το έργο των εταιριών που ε, υποβάλλουν και τις μελέτες επιπτώσεων σε σχέση με το έργο αυτό στρατηγική για παράδειγμα μελέτη επιπτώσεων αυτών των προγραμμάτων και σχεδίων. Γιατί τα λέω όλα αυτά. Εκ των υστέρων όταν έχει κάτι ε, παρουσιαστεί αντιμετωπίζουμε το θέμα των ιδιωτικών επιχειρήσεων και πρέπει να έχουμε αυτές τις μελέτες επιπτώσεων <clears throat> ώστε να μην υπάρχει ας το πω έτσι βλαπτική επιζήμια επίπτωση όταν λοιπόν υπάρχει ε, εδώ ε, συνενοχή ή συναυτουργία της εταιρείας που συντάσσει τη μελέτη επιπτώσεων και μιας μεγάλης εταιρείας για τις υποδομές σε ένα τέτοιο πρόγραμμα, ιδιαίτερα ενεργειακές εταιρείες, εταιρείες ε, που ασχολούνται είτε με ενεργειακά θέματα είτε επίσης και με ε, εκμετάλλευση ακινήτων χρειάζεται μια πάρα πολύ αυστηρή διαπίστευση ε, εταιριών που συντάσσουν αυτές τις ε, περιβαλλοντικές επιπτώσεις ώστε να είναι αντικειμενικές και αμερόληπτες. Και τέλος, αν έχουμε μια θετική γνωμοδότηση από μη κυβερνητικέ οργανώσεις, από ΜΚΟ, ΜΚΟ που κάνουν αξιόλογο, πάρα πολύ αξιόλογο έργο ε, προκειμένου να προστατευτεί η βιοπικιλότητα, ΜΚΟ που εργάζονται πανευρωπαϊκά, εγκάρσια στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Με αυτή τη συνεισφορά ε, ελπίζω ότι θα υπάρξουν τροπολογίες και είμαι πεισμένος ότι αν συνεργαστούμε με την Επιτροπή Περιβάλλοντος, ΕΝΒΗ και σε σχέση με την ε, ε, ίδια την αρμοδιότητα της ουσιοδέστερης αυτής έκθεσης θα έχουμε μεγάλη επίπτωση για να καταφέρουμε καλύτερα τα θέματα προστασίας της βιοποικιλότητας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Θα λάβει τον λόγο ο κύριος Κρέμερ τώρα, εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Παρακαλώ χωρίς μικρόφωνο. Ευχαριστώ πολύ ε, κύριε Πρόεδρο. Το έχουμε ξανασυζητήσει το θέμα αυτό, την έκθεση αυτή ε, εδώ. Εμείς ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμφωνούμε ε, με ένα τμήμα της έκθεσης, αλλά είμαστε απογοητευμένοι που δεν καταφέραμε να αντιμετωπίσουμε την μείωση της βιοπικιλότητας. Θέλουμε να συνεχίσουμε να ενισχύουμε το βασικό μέσο που έχουμε, δηλαδή την οδηγία για το οικοσύστημα και για τα πτηνά και ε, οι οποίες οδηγίες βέβαια είναι μια επιτυχία. Επίσης πρέπει να αναγνωρίσουμε τη σημασία και των οδηγιών αλλά και των ε, δικτύων που προκύπτουν από αυτές ε, και όχι μόνο τις ε, ελλείψεις των οδηγιών που αναφέρει ο εισηγητής. Ε, δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε αντιθέτως με κάποιες δηλώσεις, δηλαδή ότι υπάρχει μια χαλάρωση της εφαρμογής. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάνει ό,τι μπορεί και είναι πολλά αυτά που κάνει για να εξασφαλίσει και να ενισχύσει την εφαρμογή της οδηγίας, ειδικότερα αν δείτε τον αριθμό των παραβάσεων, ε, των διαδικασιών επί παραβάση που έχουν δρομολογηθεί για τις δύο αυτές οδηγίες, ε, είναι οι πρώτες μεταξύ όλων των διαδικασιών που έχει ξεκινήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Υπάρχουν βέβαια και κάποιες για το περιβάλλον, ε, πάνω από 400, 468 αν θυμάμαι, ε, και μόνο για το οικοσύστημα 88 ε, υποθέσεις. Υπήρξαν πολλές τέτοιου είδους διαδικασίες στο παρελθόν που έφτασαν στο δικαστήριο και δεν μιλάω μόνο για εξαιρέσεις. Έχουμε τώρα νέους στόχους για το 2020. Το Συμβούλιο ενέκρινε το Μάρτιο τα συμπεράσματά του και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι της απόψεως ότι πρέπει οπωσδήποτε τώρα να αναθεωρήσουμε, να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να επιτύχουμε τους στόχους αυτούς. Όσον αφορά τις οδηγίες, ε, συνεχίζουμε τις προσπάθειες ε, που ξεκίνησαν στο παρελθόν ειδικότερα για το δίκτυο Natura 2000 που τώρα περνά σε μια φάση διαχείρισης μετά από χρόνια κατά τη διάρκεια των οποίων ε, ε, είχαμε επικεντρωθεί στην ίδρυση, του, στη δημιουργία του, του δικτύου. Τώρα αρχίζουμε την εφαρμογή του. Εφαρμόζεται με σχέδια δράσης, με μέτρα ε, διατήρησης κλπ. Είναι και ε, σε αυτό το σημείο πολύ σημαντική η βελτίωση της συνεργασίας και του συντονισμού και στο πλαίσιο των κρατών μελών και συμφωνούμε με κάποιες από τις πτυχές της έκθεσης που αναφέρουν ότι πρέπει να ενισχύσουμε ε, την ε, δέσμευση των κρατών μελών ε, για τα δίκτυα αυτά. Πρέπει να τα ενισχύσουμε επιτόπου στα κράτη-μέλη. Αυτό δεν μπορεί να το κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχουμε ενισχύσει τις επαφές και το διάλογο με τον οικονομικό τομέα. Κάνουμε πάρα πολλά για να εξηγήσουμε την οδηγία και να πείσουμε ότι οι οδηγίες αυτές είναι ένα μέσο αηφόρου ανάπτυξης, ότι δεν έχουν σκοπό να μπλοκάρουν την οικονομική ανάπτυξη ε, και πρέπει να υπογραμμίσω ότι πολλές παρεμβάσεις αυτή τη στιγμή πιέζουν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναθεωρήσει τις οδηγίες ε, και να αποδυναμώσει ε, τον αντίκτυπό τους. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν η, ενίσχυ, η υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να πείσουμε ότι δεν παρακολύουν την οικονομική ανάπτυξη, αντιθέτως ενισχύουν την αηφόρο ανάπτυξη. Και ε, είμαστε αρκετά βέβαιοι ότι κάποιοι οικονομικοί τομείς ε, εξέφρασαν την πρόθεσή του να συζητήσουν με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να μην υπάρξουν ε, συγκρούσει και να συνεχίσουμε την επίτευξη του στόχου της διατήρησης βιοποικιλότητας στο πλαίσιο της αηφόρου οικονομική ανάπτυξη. Αναφερθήκατε ε, και σε κάποια άλλα ζητήματα που είναι σημαντικά, για συνοριακή συνεργασία για παράδειγμα. Και από αυτού όμως τα κράτη-μέλη είναι υπεύθυνα προκειμένου ε, τα, να συνεργάζονται με τους γειτονές τους για να υπάρχει μια συνοχή του δικτύου Natura 2000 γιατί η βιοπικιλότητα δεν ε, είναι δυνατόν ε, να ε, διατηρηθεί μόνο σε πολύ συγκεκριμένα σημεία. Πρέπει να υπάρχει μια συνοχή, να μην διασπάται πουθενά η αλυσίδα και πρέπει να υπάρχουν και εθνικά συμπληρωματικά δίκτυα και οριζόντιες πολιτικές ε, διατήρησης των ειδών ε, που να ισχύουν σε ολόκληρη την επικράτεια. Εμείς προσπαθούμε λοιπόν να συνεργαστούμε με τα κράτη-μέλη για να εξασφαλίσουμε την συνοχή αυτή του δικτύου. Θα ήθελα επίση να υπενθυμίσω τέλος ε, ότι έχουμε μια νέα ομάδα επιρογνωμόνων με, με τα κράτη-μέλη και τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις για να συζητήσουμε τη διαχείριση του Natura 2000 και να βελτιώσουμε τη συνοχή του και τη διαχείρισή του στο μέλλον. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πέρυσι παρουσίασε μια ανακοίνωση για την οδηγία εκτίμησης ε, περιβαλλοντικών ε, επιπτώσεων ε, και είδαμε τι περιθώρια υπάρχουν βελτίωση, βελτίωσης της. Τώρα για τους χρόνους αντίδρασης, το αναφέρατε επίση. Κοιτάξτε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπαθεί να απαντήσει το συντομότερο δυνατόν για τις αναφορές ε, ε, και τις ε, τις διάφορες ε, προσφυγές, όμως δεν μπορούμε να ξεκινήσουμε διαδικασία επί παραβάση όταν δεν υπάρχει ακόμη παράβαση, όταν δεν έχει διαπιστωθεί παράβαση. Έχουμε όμως διαδικασίες όπως για παράδειγμα το πρόγραμμα ε, το πιλωτικό συνεργασίας με τα κράτη-μέλη για την διαχείριση ε, των προσφυγών. Αυτό έχει ήδη επιφέρει κάποια θετικά αποτελέσματα. Αυτά. Μακρηγόρησα, οπότε θα σταματήσω. Σας ευχαριστώ. Ξεκινάει η συζήτηση. Okay. I'll do in English this time. Αγγλικά αυτή τη φορά. Έχω την εντύπωση ότι είχαμε θέμα μεταφραστικό την τελευταία φορά όταν είχαμε δανέζικα τα οποία χρησιμοποιούσαμε. Ίσως έτσι θα μπορέσει να σχολιαστεί άμεσα αυτό το θέμα με τη συμπαρέμβασή μου. Θέλω και πάλι να ευχαριστήσω πολύ για την έκθεση αυτή. Και υπάρχουν πολλά σημαντικά πράγματα. Επίσης ε, και προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ευχαριστώ εξακολουθούμε να υφιστάμεθα τα αρνητικά στα κράτη-μέλη και στη δική μου χώρα σε σχέση με αυτή την οδηγία. Σαν να ήταν απλά και μόνο κάποιες καλές συμβουλές και όχι κανονισμοί και κανόνες. Θα ήθελα εδώ να προσθέσω ότι κάθε φορά όταν έχουμε μια διαδικασία παραβίασης ή επιπαραβάση είναι και κλεισμένο των θυρών. Δεν μπορούμε να παραστούμε. Είναι πολύ κακό αυτό για το έργο και στα Εθνικά Κοινοβούλια να μπορεί να παρακολουθήσει τι γίνεται εδώ. Μπορώ να παρακολουθήσω υποθέσεις στη Δανία όπου η κόρη μου είναι πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος εκεί στο Κοινοβούλιο και δεν μπορούν να δώσουν συνέχεια και να παραστούν. Και θα ήθελα να πω θα έπρεπε με αυτό να ασχοληθούμε κι εμείς και θα ήθελα να ζητήσω, να ρωτήσω μήπως θα έπρεπε τις συστάσεις αυτές από την WWF, το Ταμείο για την Προστασία της Φύσης, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε και να εξετάσουμε τις προοπτικές. Έχουμε και ηλεκτρονικό μήνυμα, είναι νομίζω πολύ συνετές οι σύμβουλες που μας δίνουν. Και θα μπορούσα επίσης να ζητήσω για να αποσαφινιστεί αυτό, να έχουμε συγκεκριμένα χειροπιαστά παραδείγματα κάτι για παράδειγμα και από την Δανία για την ε, ε, δράση αυτή. Έχοντας παραδείγματα λοιπόν θα μπορούμε να προχωρήσουμε. Τώρα για την πιο χαλαρή συνέχεια που δίνεται για την οδηγία για την προστασία της φύσης. Πιστεύω ότι ακόμα και όταν ακούμε τον κύριο Μπαρόζο, τουλάχιστον όταν ήταν στην ομάδα μου και μας μιλούσε, κάνοντας ε, λόγο για την αναθεώρηση αυτής της οδηγίας, αποκομίσαμε την εντύπωση ότι αυτή η προσαρμογή θα κάνει τα πράγματα πιο εύκολα στην χειροπιαστή εφαρμογή. Δεν είναι θέμα τώρα οδηγιών εδώ, αλλά σεβασμού και συμμόρφωσης με αυτές τις συστάσεις και οδηγίες. Γι' αυτό πρέπει να λάβουμε υπόψη αυτό το οποίο συνιστά η WWF η κυρία και ο Αλίστερ Τέιλορ. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Μάια, ευχαριστώ Πρόεδρε. Εγώ χαιρετίζω την έκθεση, την γνωμοδότηση του κυρίου Μποστινάρου για το επίπεδο των απαιτήσεων και διεκδικήσεων. Σημερίζομαι απόλυτα αυτές τις απαιτήσει σε σχέση με την ανάγκη προστασίας της βιοπικιλότητας σίγουρα, κατανοώντας ότι δεν έχει σύνορα η βιοπικιλότητα και συμμερίζομαι αυτές τις απαιτήσεις, διότι η διάγνωση για την μητέρα γη δεν θα μπορούσε να είναι αρνητικότερη. Η πάντσα μάμα, πως την αποκαλούν οι Ινδιάνοι, βρίσκεται σήμερα κατάκητη. Δεν είναι λοιπόν ένα θέμα ίσονος σημασίας. Έχουν πολύ μεγάλη ευθύνη τα κράτη-μέλη. Αυτό το οποίο διακυβεύεται και κινδυνεύει είναι η ίδια η ζωή, η ζωή υπό ευρύτερη έννοια, η ίδια η επιβίωση των ανθρώπινων όντων. Στην Κοπερχάγη ήταν σχεδόν αναπόφευκτο θεωρούσαμε στο να καταλήξουμε σε μια αύξηση ε, θε, της θερμοκρασίας του πλανήτη στους 2,5 βαθμούς Κελσίου και είναι σαφές ότι αν καταλήξουμε σε αυτήν την αύξηση 2,5 βαθμών ε, ε, Κελσίου κατά μέσον όρων τότε θα ε, κινδυνεύει η επιβίωση και γι' αυτό έχουμε μεγάλη ευθύνη οι χώρες εκείνες που παραγούν μεγαλύτερη ποσότητα διοξιδίου του άνθρακα και θερμοκηπίων του αερίου γι' αυτό αυτές οι απαιτήσει πρέπει να είναι πολύ πιο αυστηρές σε πολύ υψηλότερο επίπεδο. Νομίζω η γνωμοδότησή μας στοχεύει στη σωστή κατεύθυνση. Πρέπει να είμαστε πολύ πιο απαιτητικοί με εμάς τους ίδιους για να δώσουμε παράδειγμα, υποδειγματικά να δράσουμε ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι υποδειγματική σε παγκόσμια κλίμακα για την βιοπικιλότητα. Αν δεσμευθούν όλες οι ήπειροι με αυτές τις αυστηρές ε, απαιτήσει για να αντιμετωπιστεί ο κίνδυνος που αντιμετωπίζει η ζωή, τότε μπορούμε να επιβραδύνουμε αυτές εξελίξεις ξεκινώντας μια πορεία προς μια αυθεντική προστασία και προάσπιση της βιοπικιλότητας. Γι' αυτό συμμερίζομαι αυτό το επίπεδο αυστηρών απαιτήσεων και θα συμμεριστεί η ομάδα μου αυτές τις αρχές κύριε Μποστινάρου για να μπορέσουμε να έχουμε μια διεργασία ώστε που, μια και έχουμε θέμα που ξεπερνά τα σύνορα είναι διασυνοριακό να μπορέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να δώσει το υπόδειγμα, το παράδειγμα στο σεβασμό στην ευθυγράμμιση για τη διασφάλιση της αηφορίας και της βιοπικιλότητας. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Σα Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ και τον κύριο εισηγητή Μποστινάρο για την έκθεσή του. Θα έλεγα τρία προβλήματα τα οποία υφίστανται, τα αναφέρει σωστά, θα μας απασχολήσουν και πρέπει αντίστοιχα να διατυπώσουμε τροπολογίες για να εμβαθύνουμε στα θέματα αυτά. Ο στόχος είναι σαφής και τον στόχο τον δέχονται όλοι και παντού αναφέρεται θα έλεγα σε όλους τους λόγους που εξτομούμε όλοι είμαστε υπέρ όλοι είμαστε υπέρ της προάσπισης της βιοπικιλότητας να μην επιδεινωθεί η κατάσταση να διατηρηθεί η βιοπικιλότητα καλά μαντάτα αυτά αν ειμαστε ειλικρινεί, ειλικρινείς υπάρχει όμως εδώ ένα πρόβλημα πολλά κράτη-μέλη αντιμετωπίζουν τους νόμους, τα νομοθετήματα και τους κανονισμούς ως εμπόδια στις επενδύσεις και αντιδρούν και μάλιστα προσβάλλονται όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση ή η Επιτροπή Αναφορών στρέφονται στα κράτη-μέλη και λένε στο κράτος μέλος ή στα κάποια κράτη-μέλη εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα, μπορείτε να μας δώσετε μια έκθεση και να αναφερθείτε σε αυτό. Είναι ένα θέμα στο οποίο υποστηρίζω ρητά τον εισηγητή. Χρειαζόμαστε προθεσμίες και διορίες για αυτόν τον διάλογο. Με την καλή έννοια, διότι αν σε μια διαδικαστική υπόθεση συζητά κανείς θέματα, τότε μπορεί κανείς προβλήματα να τα σταθμίσει και να τα αξιολογήσει και να τα άρει, να τα αντιμετωπίσει σωστά. Για ένα τέτοιο διάλογο χρειαζόμαστε διορίες και προθεσμίε. και είναι πολύ σημαντικό και χρειαζόμαστε και κριτήρια όταν εμείς, και αυτό είναι το δεύτερο θέμα και υποστηρίζω και σε αυτό τον εισηγητή, όταν και αν εμείς πραγματικά σοβαρέ ελλείψει και ελλείμματα διαπιστώνουμε, τότε θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναλαμβάνει δράση. Δεν έχει κανένα νόημα αν κάποιο τέτοιο εγχείρημα, για παράδειγμα, μέσω μη διαλόγου δεν προχωράμε, παγώνουν, σταματούν τα πράγματα, τότε στενεύουν τα περιθώρια, λίγουν οι δυνατότητες, η βιοπικιλότητα ούτως ή άλλως βλάπτεται και υφίσταται ζημιές. Δεν θα έπρεπε να είχε δοθεί μια τέτοια έγκριση για ένα τέτοιο πρόγραμμα και τι θα κάνουμε τώρα εκ των υστέρων και έρχονται κάποιοι και λένε εντάξει πρέπει να υπάρξουν αντισταθμιστικά μέτρα. Καλύτερο είναι μέσα σε μια διαδικασία τακτή να συζητά κανεί. και διορίε και προθεσμίε είναι σημαντική υπόθεση. Με μεγάλε παραβιάσει και παραβάσει πρέπει κανεί να είναι αυστηρό. Τώρα εδώ σε σχέση με το επόμενο θέμα διτά πρέπει να το δούμε. Δεν έχει αναπτυχθεί επαρκώ. πρώτο σημείο συνεργασία Ευρωπαϊκή Ένωση και εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση χωρών. Και αυτό σημαντικό. Και μέσα στην ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν μεγάλε ελλείψεις και ελαττώματα. Έχω κάμια φορά την εντύπωση ότι υπάρχουν κράτη-μέλη που προγράμματα επενδύσεων να εντάσσουν στις ε, μεθοριακές περιοχές και μετά άλλη χώρα, γειτονική χώρα, παραπονείται ότι δεν έχει εμπλακεί επαρκώ, Χρειαζόμαστε κανόνε για την προστασία του περιβάλλοντο. διότι η βιοπικιλότητα δεν σταματά στα σύνορα. Συμφωνώ λοιπόν με αυτά τα τρία σημεία που αναφέρατε κύριε Μποστινάρου. Είναι πολύ σημαντικά διασυνορική συνεργασία, προθεσμίε και διορίε και αυστηρά κριτήρια. Και αν καταφέρναμε στο τέλος τέλος να είχαμε, πώς να το πω, να διασφαλίσουμε την ύπαρξη της βιοπικιλότητας, τη διατήρησή της ή να το κατανοήσουν ως ευκαιρία αυτό τα κράτη-μέλη και όχι ως εμπόδιο για επενδύσεις θα είχαμε σημειώσει μια μεγάλη νίκη αλλά πόρο απέχουμε από αυτήν ακόμα. Κανείς άλλος δεν επίθυμει το λόγο. Ο εισηγητής Μποστινάρο έχει το λόγο. Σάπτε στα Ιταλικά η απάντηση. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι ένας από τους λόγους ύπαρξης έκθεσης μου είναι η έκθεση του κυρίου Ιτουργκάης ο οποίος με πάρα πολύ σοβαρά επιχειρηματά έδειξε ότι η περιφαλοντική πτυχή είναι μεταξύ των σημαντικότερων ε, από την άποψη των Ευρωπαίων πολιτών. Οι περισσότερες αναφορές έχουν να κάνουν ε, με το ζήτημα της παραβίασης των περιβαλλοντικών κανόνων και την εφαρμογή των ε, ευρωπαϊκών προτύπων. Όσον αφορά τώρα τις παρατηρήσεις ε, του εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θα ήθελα να πω τα εξής. Πρώτον, είναι γεγονός ότι το περιεχόμενο της οδηγίας πάντοτε καλό είναι. Και εγώ δεν αμφιβάλλω καθόλου ε, γι' αυτό δεν προτείνω να το αναθεωρήσουμε το περιεχόμενο, να το αλλάξουμε. Το βασικό πρόβλημα είναι η εφαρμογή και η έκθεση μου αγωνίζεται για αποτελεσματική εφαρμογή των οδηγιών είτε που αφορούν ε, τη βιοπικιλότητα είτε το δίκτυο Natura 2000. Και επίσης ε, αφορά την εφαρμογή. Όσον αφορά τις σχέσεις, μιλήσατε για τις σχέσεις ε, μεταξύ των ε, χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών που δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τους ή άλλως έχουμε ήδη συμφωνίες νομικής φύσεως, είτε η στρατηγική σχέση συνεργασίας με Ευρωπαϊκής μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ρωσίας, για παράδειγμα, ή Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ουκρανίας, Ευρωπαϊκής Ένωσης και Μολδαβίας υπάρχουν ε, τέτοιου είδους ε, συμφωνίες με τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων ανεξαρτήτως με το αν είναι υποψήφιες χώρες ε, ή χώρες που θα συμπεριληφθούν στον κατάλογο των χωρών που θα προσχωρήσουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε συγκεκριμένους νομικούς κανόνες, έχουμε διμερεί μέσα ή πολυμερή ε, μερικές φορές, αλλά πρέπει οπωσδήποτε το ζήτημα, τα ζητήματα αυτά ε, της προστασίας της βιοπικιλότητας ε, πρέπει να τα συμπεριλάβουμε στις συμφωνίες μας με τις χώρες αυτές. Εύκολο είναι να κατηγορούμε και επιμένω στο σχέδιο North Stream. Η Ρωσία υπέγραψε τη σύμβαση ΕΣΠΟ αλλά ποτέ δεν την επικύρωσε, δεν την έχει, επικυρώσει, δεν την έχει επικυρώσει τη σύμβαση αυτή. Είναι γεγονός ότι δεν υπάρχει καμία αναφορά στο θέμα αυτό της αναγκαιότητας της επικύρωσης της ε, σύμβασης αυτής δεν γίνεται καμία αναφορά στις σχέσεις, στις συνομιλίες Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη Ρωσία για αυτό το θέμα. Ε, και ούτως ή άλλως το θέμα αυτό θα μας απασχολήσει άμεσα γιατί άρχισε η κατασκευή το 2010. Πώς λοιπόν θα προστατεύσουμε τη βιοπικιλότητά μας αν μας λείπουν, μας λείπουν τα σημαντικότερα νομικά μέσα. Αυτό είναι αποστολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περισσότερο από ε, αποστολή των κρατών μελών. Και τρίτον, ε, έχουμε χώρες ε, όπως για παράδειγμα οι χώρες του Μαγκρέμπ και έχουμε και την ένωση τους. Πρόκειται για μία ε, συγκεκριμένη σχέση που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση με τις χώρες ε, Μαγκρέμπ. Για ποιο λόγο να μην ε, εισαγάγουμε προοδευτικά μετά από διαπραγμάτευση και μετά από διάλογο να κινηθούμε προς αυτή την κατεύθυνση, να τη συμπεριλάβουμε, να συμπεριλάβουμε τα πρότυπα αυτά και σε αυτές τις συμφωνίες. Να μην διαπιστώνουμε απλώς το μοιραίο του πράγματος όταν φτάνουμε στο μη περαιτέρω. Αφού τα γνωρίζουμε ήδη όλα αυτά. Αυτή είναι η δική μου ανησυχία. Και όσον αφορά τώρα τα σχόλια της κυρίας ε, Όκιν, θα ήθελα πάρα πολύ να σας ευχαριστήσω για την υποστήριξή σας. Συμφωνώ απολύτως με όσα είπατε για την ε, ε, συνεισφορά της ΒΒΕΦ Έχουμε πάρα πολλές αναφορές από όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν είναι δυνατόν να αναφερόμαστε όμως σε κάθε αναφορά. Τότε αντί για τρεις σελίδες ε, θα έχουμε ολόκληρη βίβλο παραβίασης των ευρωπαϊκών κανόνων και κανονισμών για την βιοπικιλότητα. Γνωρίζουμε πολύ καλά ε, στο πλαίσιο της Επιτροπής μας η περιβαλλοντική πτυχή είναι από τις σημαντικότερες Όσον αφορά τώρα αυτά που είπε ο κύριο Γιάρ, συμφωνώ ότι είναι ένα πρόβλημα εφαρμογής ε, και από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής και από πλευράς ε, κρατών μελών πολλά πρέπει να γίνουν για να βελτιωθεί η εφαρμογή και βέβαια υπάρχει ανάγκη διαλόγου, να υπάρχει ένας σοβαρός διάλογος και θα ήθελα να ευχαριστήσω ε, όλους τους συναδέλφους για την ε, συμβολή τους και θα ήθελα να επιμείνω στη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να επιτύχουμε το καλύτερο δυνατό μέσο για να ε, προστατεύσουμε τη βιοπικιλότητά μας. Ευχαριστώ πολύ. Να ευχαριστήσω τον συνάδελφο Μποστινάρου. Δεν ξέρουμε ακόμα το χρονοδιάγραμμα των εργασιών Λοιπόν, μάλλον το Σεπτέμβριο θα μπορούσαμε να ορίσουμε λοιπόν και την προθεσμία για τις Ίσως να το κάνουμε την επόμενη φορά και μέσω email θα σας γνωστοποιήσουμε αυτή την ομοιρημηνία για, πριν, για τη συζήτηση σε τελική φάση. Το επόμενο σημείο τώρα είναι το σημείο 21. 1098 του 2007 ο αναφέρον είναι απόν. Ο Πίτερ Βάιντερ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αυτή η αναφορά αφορά την, <clears throat> το διελιστήριο πετρελαίου Σαν Ρόκε στο Γιβραλτάρ, Σρέψα και θα ήθελα να αναφερθώ σε δύο ε, ε, έρευνες από τη ΒΙΤΟ, το Φλαμανδικό Ίδρυμα Περιβαλλοντικών Μετελών, Μελετών, η άλλη από την ΆΙΣΙΑ, την Ένωση για την, ε, τις έρευνες ε, της βιομηχανικής συνεργασίας στην Ανδαλουσία. μετά μία μελέτη όσον αφορά την εγκατάσταση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με, τις, ε, με τον σύμβουλο ΕΝΤΕΚ. E Όλες αυτές οι εκθέσεις επιβεβαιώνουν ότι οι επιδόσεις του δηληστηρίου βρίσκονται κοντά στις καλύτερες επιδόσεις ε, τεχνολογικά που περιγράφονται σε σχέση με την, την οδηγία ενσωμάτωσης ε, της, του ελέγχου της περιβαλλοντικής ρήπανσης Ωστόσο όμως υπάρχει περιθώριο για βελτιώσεις. Σαν αποτέλεσμα λοιπόν αυτών των μελετών προληπτικά μέτρα προτάθηκαν να ληφθούν και υπήρξε ένα διευρυμένο πλαίσιο. Τα συμπεράσματα της μελέτης ε, εντάχθηκαν και εγγράφησαν στην αδειοδότηση της εταιρείας ένα πρόγραμμα δράσης ε, επίσης ε, προβλέφθηκε σε σχέση με τις εγκαταστάσεις. Θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι αυτά τα δύο τελευταία μέτρα, η συμπερίληψη στην αδειοδότηση και το πρόγραμμα δράσης από πλευράς της εκμεταλλεύτριας εταιρείας θα πρέπει σε σχέση με τις αρχές να, να επακούν. Καμία άλλη δράση δεν μπορεί να, να αναλυθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτή τη στιγμή. Επιπλέον θα ήθελα να επισημάνω και κάτι άλλο, ότι μια διαδικασία παραβάση είχε ξεκινήσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με βάση την παραβίαση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα της ατμόσφαιρας όσον αφορά την νομοθεσία σε σχέση με την Οδηγία 99 κάθετος 30 επίσημη γνωστοποίηση απεστάλη τον Ιανουάριο 2009 προς την ε, Ισπανία και μια αιτιολογημένη <clears throat> γνωμοδότηση ε, υποβλήθηκε τον Μάρτιο. Ωστόσο όμως ε, δεν αφοράται πλέον η ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα στο Γιβρατά διότι οι προδιαγραφές ευθυγραμμίζονται σε σχέση με το 2008 και τα προσωρινά στοιχεία επίσης δείχνουν συμμόρφωση και για το 2009 όσον αφορά την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα στο Γιβραλτάρ. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε για την ενημέρωση και ο συνάδελφος Μάγερ έχει το λόγο. Ευχαριστώ, ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω τους αναφέροντες ε, που για τις προσπάθειές τους σε μία αναφορά και από την Ισπανία και από το Γιβραλτάρ, από το Ηνωμένο Βασίλειο. Ζητούν όλοι και λένε ότι θα πρέπει να γίνει μια επιδημιολογική έρευνα από τη στιγμή που υπάρχει ένας κίνδυνος κοινωνικός. Το ίδιο και στην Βέλβα σε μια πρόσφατη επίσκεψή μας όταν ακούσαμε από διάφορους σημαντικούς στην Ισπανία όπως ε, σχετικό Ιστιτούτο που δείχνει τη θνησιμότητα από καρκίνο στην Ισπανία και στο Καντίθ ε, και στην περιοχή του Γιβραλτάρ είναι η θνησιμότητα από τις υψηλότερες όσον αφορά τον καρκίνο. και από το Πανεπιστήμιο Φάμπρα της Βαρκελόνης που επικυρώνει, επιβεβαιώνει αυτά τα στοιχεία είναι πάνω από τη μέση εθνική εθνισιμότητα, λευχαιμίες πνευμόνων, στομάχου κλπ. κλπ. Η επιστημονική κοινότητα παρόλα αυτά δεν έχει μελετήσει όπως πρέπει. Μας το είπαν αυτό στη Βέλβα τι γίνεται για την μόλυνση εκεί δεν μελέτησαν όπως πρέπει επιστημονικά, δεν υπάρχουν βεβαιότητες προς το παρόν εάν αυτοί οι θάνατοι προέρχονται από μια ορισμένη βιομηχανική δραστηριότητα συγκεκριμένη. Δεν υπάρχει λοιπόν σιγουριά. Και η αναφορά βέβαια είναι πολύ λογική. Όταν θα ασχοληθούμε με τη Βέλβα και ελπίζω, εύχομαι ότι θα μπορούσαμε να συστήσουμε στις αρχές ε, όλες αυτές οι μελέτες να γίνουν με συντονισμένο τρόπο ώστε να μπορέσουμε επιστημονικά να έχουμε μια επιδηλωμελογική έρευνα και αποτελέσματα, πορίσματα και να δούμε πού οφείλεται αυτή η υψηλή θνησιμότητα πάνω από την μέση εθνική παρόμοια. Και αυτά που οφειλεται αυτη η ψηλη θνησιμοτητα πανω απο την μεση εθνικη παρομοια και αυτα που συμβαινουν στη Βέλβα, τι γίνεται από την ακτινοβολία, από σκόνες, στάχτες κλπ. Τι ακριβώς, από πού συμβαίνει, από πού σε τι οφείλεται και στο Γιβραλτάρ. Νομίζω ότι αυτή η επιδημιολογική έρευνα θα μπορούσε, πρέπει να μας βοηθήσει για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το σχετικό πρόβλημα με αυτή την υψηλή θνησιμότητα σε σχέση με το εθνικό επίπεδο. Αυτά είναι και κοινή λογική βέβαια και αυτό μπορεί να κάνει εδώ η Επιτροπή μας είναι μια επιστολή να απευθύνει, να πει ότι έλαβε την αναφορά αυτή και ότι θα προχωρούσαμε σε συστάσεις για την επιδημιολογική έρευνα. Οι αρμοδιότητες είναι εθνικές και όχι βέβαια ε, κοινοτικέ. Εντάξει, αλλά οι συστάσει δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι και καλά μόνο εθνικέ. Σύσταση είναι, μπορεί να είναι και τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα λοιπόν και στο Γιβραλτάρ και στην Ισπανία και στην ε, Ηνωμένο Βασίλειο να εργαστούν από κοινού οι επιστήμονες, να συνεργαστούν για να μπορέσουν να καθησυχάσουν τον κόσμο και αν όμως ε, αποδειχθεί ότι λόγω αυτής της δραστηριότητας αυτή προκαλεί ε, παρόμοιες ασθένειες, ε, τότε θα πρέπει ε, από την Εκκλησική Επιτροπή να υπάρξει κάτι, να γίνει κάτι, να ξεκινήσει η επίσημη εξέταση του θέματος και να μπορέσουμε έτσι να βοηθήσουμε πάντως με τη σχετική σύσταση για την επιδημιολογική έρευνα. Αυτά. Η Πρόεδρος. Καμία άλλη παρέμβαση. Όχι τότε... Αυτό που ακούσαμε από τον συνάδελφο Μάγερ θα μπορούσαν να γίνουν δεκτά, δηλαδή να απευθύνουμε μια επιστολή στις αρμόδιες αρχές και να δούμε και συμπληρωματικά μια σύσταση πώς μπορούμε να απευθύνουμε, μπορεί να γίνει αυτό και να υπάρξει μια μελέτη, να δούμε, να επιβεβαιώσουμε τις μελέτες που είναι στη βάση αυτής της αναφοράς θα μπορούσαμε να το κάνουμε αυτό λοιπόν, ταυτόχρονα όμως γοργά να προχωρήσει η αδικασία γιατί καταλαβαίνουμε ότι θα υπάρχουν δραματικές συνέπειες αν όλα αυτά αληθεύουν. Παραμένει ανοιχτό το θέμα λοιπόν, έτσι και θα προχωρήσουμε. Προχωράμε παρακάτω, είναι 22 αναφορά 439-2009 της κυρίας Έλσα Αϊμόνα Ιταλικής Ιθαγένειας και Αντώνη Μονσερά έχει το λόγο από την Επιτροπή. Ευχαριστώ πολύ. Ε, πρόκειται για την κίστη του Ταρλόφ, ε, που είναι μία μειοσκελετική διαταραχή και είναι πηγή ε, πολλών προβλημάτων. Υποφέρουν πάρα πολλοί πάρα πολύ από αυτό το ζήτημα. 6.000, με τη μεταξύ των 6.000 ε, ε, ε, σπάνιων ασθενειών είναι ένα από τα βασικά προβλήματα δημόσιας υγείας μεταξύ 24 και 30.000 Ευρωπαίων, δηλαδή 6 8% του ευρωπαϊκού πληθυσμού υποφέρουν από αυτήν. υπήρξε μια σύσταση του Συμβουλίου για το θέμα αυτό υπό την Τσεχική Προεδρία τον Ιούνιο του 2009 αυτό που δεν έχει σκοπό να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί ούτε οικονομικό το μπορεί, ούτε πολιτικό το μπορεί, είναι να υπάρξει μια εξατομικευμένη πολιτική για, μια, για κάθε μία από τις 6.000 σπάνιες ασθένειε. Θα υπάρξει μια ολοκληρωμένη ε, προσέγγιση για το θέμα των ε, σπανίων ασθενειών και η ανακοίνωση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και, και η σύσταση του ε, Συμβουλίου προτείνουν κάποια μέσα επιστημονικού ε, και κλινικού χαρακτήρα που πρέπει οπωσδήποτε να εφαρμοστούν για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα αυτά, είτε δίκτυα να υπάρξουν, είτε βελτίωση στα, ε, πρόσβαση στα ορφανά ε, φάρμακα, βελτίωση της καταχώρησης και ταξινόμησης των σπανίων ασθενειών, και ειδικότερα για την περίπτωση της κίστης ε, Ταρλόφ ε, είναι γεγονός ότι κάποιες χώρες, ε, ειδικότερα η Γαλλία, δεν την θεωρούσαν σπάνια ασθένεια παρά το γεγονός ότι είναι ένα ζήτημα που επηρεάζει ένα κομμάτι του ε, πληθυσμού της Γαλλίας. Ε, είναι πέντε στους 10.000 ε, υποφέρουν από αυτήν. Δηλαδή από απόψε ως εμφάνιση συχνότητας τα ποσοστά είναι πολύ χαμηλά. Επιμείναμε στο πλαίσιο της βάσης δεδομένων για τα, τις σπάνιες ασθένειες να συμπεριληφθεί και η κίστη αυτή ε, και έγινε αυτό το Φεβρουάριο του... Ε, για να συμπεριληφθεί και αυτό το καταφέραμε το Φεβρουάριο του 2010. Ε, θα συμμετάσχουμε σε μία, συνεδρί... σε μία συνάντηση στο Σαμπερί και αυτό είναι κάτι που δεν έχει ε, συμβεί ξανά στο παρελθόν ε, και θα δούμε πώς μπορούμε να οργανώσουμε μία πρωτοβουλία για να ευαισθητοποιήσουμε, να γίνει πιο γνωστή των, ε, πιο γνωστές οι πτυχές αυτής της ασθένειας. Τα κοινοτικά προγράμματα μας το επιτρέπουν να το κάνουμε αυτό. Υπάρχουν πολλά προγράμματα σπανίων ασθενειών ε, τα οποία έχουμε υποστηρίξει, αλλά το να υπάρξει ένα νέο δίκτυο, ε, όπως για παράδειγμα ε, για το πρόβλημα της κίστης Ταρλόφ, είναι κάτι το εντελώ καινούριο. Επειδή έχει ξεκινήσει όλη η διαδικασία από τις 19 Μαρτίου του 2010, ελπίζουμε ότι εντός του 2011 θα ξεκινήσει το δίκτυο αυτό. Έχουμε προσπαθήσει να συμπεριλάβουμε σε αυτό το δίκτυο όλα τα προγράμματα σπανίων ασθενειών που πληρούν βέβαια τα απαραίτητα ε, κριτήρια. Γνωρίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή της μεγάλης δυσκολίας ε, που δημιουργεί αυτή η ασθένεια και είναι και πολύ ιδιαίτερο ε, το θέμα και υπάρχουν πολύ, υπάρχει πολύ λίγη εμπειρογνωμοσύνη είναι πολύ για αυτή την σπάνη ασθένεια. οι γνώσεις, πολύ ασθενών. Αλλά είναι γεγονό ότι οι ερευνε για αυτήν τη σπάνια ασθένεια, κάτι που περιπλέκει ακόμη περισσότερο τη ζωή των ασθενών. Αλλά είναι γεγονο ότι η ασθένεια αυτή, στο πλαίσιο της, ε, των πρωτοβουλειών τη ευρωπαικη επιτροπη για τι σπάνιες ασθένειε αποτελούσε και εξακολουθεί να αποτελεί προτεραιότητα. Θα ήθελα να σα ευχαριστήσω. Το σημειώνω ότι η Επιτροπή δείχνει μια ευαισθητοποίηση για το θέμα, αλλά παρακαλώ διευκρινίστε μου κάτι λέτε ότι ξεκίνησε μια διαδικασία ώστε αυτή η περίπτωση να συμπεριληφθεί στις σπάνιες ασθένειες ή μήπω απλά και μόνο θα πρέπει να ενεργοποιηθεί, από ποιον θα πρέπει να ενεργοποιηθεί αυτή η διαδικασία για να ενταχθεί στις σπάνιες ασθένειες. Για πέστε μου. Η διαδικασία έχει κλείσει η Επιτροπή θα πρέπει να έχει ζητήσει από την Orphanet είναι η επίσημη βάση στοιχείων για περίπου 6.000 σπάνιες ασθένειες και εκεί να τρέχουν οι επαγγελματίες του κλάδου για να ξέρουν ποια είναι, τι χαρακτηριστικά έχει μια σπάνια ασθένεια. Ε, γιατί κανείς γιατρός δεν μπορεί, εκτός από τον Δόκτωρα Χάους την τηλεοπτική σειρά, κανείς άλλος δεν αναγνωρίζει τη φύση μιας ε, σπάνιας ασθένειας εύκολα. Άρα λοιπόν ανατρέχουν σε αυτή την ορφανέτ για να δούνε τα χαρακτηριστικά τους κλπ. Και μέχρι το 2009 είχαν αρνηθεί εκεί την Κίστη Τάρλοφ να τη συμπεριλάβουν. Εμείς ε, επιμείναμε επιστημονικά συζητώντας και λοιπά. Τελικά έγινε δεκτή και τώρα η Κίστη Τάρλοφ όλα αυτά είναι στη βάση στοιχείων Orphanet. Λοιπόν, ε, νομίζω ότι η Επιτροπή μισκάναμε κάναμε ό,τι έπρεπε να γίνει. Ευχαριστώ. Εντάξει, λέει η πρόεδρος. θα μπορούσε να κλείσει η αναφορά αυτή γιατί έκανε ό,τι έπρεπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της. Καμία αντίρρηση. Όχι. Τότε εντάξει. Στους αναφέροντες ε, θα, στους αναφέροντες θα τους ενημερώσουμε. Πάμε τώρα στην 27. Ρομπέρτο Τζουραστάντε, Ιταλικής Ιθαγένειας, σχετικά με τη ρήπανση. Και τώρα δεκαστήλιο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Αφορά την αποκατάσταση μιας περιοχής μπαζώματος. Αυτή η χωματερία έκλεισε το 1993 και σύμφωνα με τον αναφέροντα μεγάλος κατάλογος θεμάτων μόλυνσης του περιβάλλοντος πρέπει να διερευνηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επτά θέματα υπάρχουν, θα τα απαριθμίσω αυτά. Πρώτον, διοξίνες στο έδαφος. Μετά από έρευνες που έγιναν από την Επιτροπή μαζί με τις αρμόδιες αρχές, πήραμε πληροφορίες από ένα δημόσιο ε, πειραματικό εργαστήριο. Σύμφωνα με αυτές τις πληροφορίες δεν είχε εντοπιστεί πρόβλημα επ' αυτού ακόμα. Δεύτερον, στάχτη, τέφρα που εκτίθεται, μια και η χωματερή είχε αποτέφρωση και είχε στοιχεία τεφρών και έτσι αυτές αποκαλύφθηκαν και υπήρχαν προβλήματα και με διοξίνες. Αυτό το θέμα επανορθώθηκε έχοντας διαστρωμάτωση ε, ε, ε, και έχουμε επίσης και το θέμα του αμοιάντου. Επίσης σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε δεν βρέθηκε, δεν είναι βάσιμη η κατηγορία για την ύπαρξη αμοιάντου. Τέταρτον, ε, μόλυνση των υπεδαφίων υδάτων. Πάλι αυτό δεν ε, ε, θεωρείται βάσιμη κατηγορία από την έκθεση. Μετά, μόλυνση σε σχέση με το θαλάσσιο είδο, το θαλάσσιο νερό. Ούτε και αυτό επιβεβαιώθηκε. Και εδώ έχουμε δύο σημεία από των οποία χρειάζονται έρευνε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά το έδαφος το οποίο έχει λέει, υποστεί ε, τη μέσα ρήπανσης πάνω από τα κατόφλια και μετά όσον αφορά την μόλυνση του ε, πυθμένα της θάλασσας. Εδώ υπάρχει λοιπόν ένας, μια τεράστια απαρίθμηση από πλευράς του ε, συντάκτη. Όλα όσα βρίσκονται σε αυτή τη χωματερή έχουν υποστεί λέγεται αυτές τις βλάβες. Ήρθαμε σε επαφή με τις αρμόδιες αρχές, τις Ιταλικές αρμόδιες αρχές για να διακριβώσουμε το θέμα αυτό και σε μια επιστολή που λάβαμε πέρσι ανέφεραν οι Ιταλικές αρχές στο σημείο υπαριθμών 1 δηλαδή σε σχέση με τα εδάφη που ξεπερνούν τις τιμές κατόφλια λένε ότι περιορίζεται η μόλυνση σε σχέση με τις όχθες και ότι δεν υπάρχει υπέρβαση που να θέτει σε κίνδυνο είτε ανθρώπους είτε ε, την θαλάσσια περιοχή. Δεύτερο σημείο για τα, τον πυθμένα της ε, θάλασσας ε, και τα ειζήματα του πυθμένα με μόλυνση από διοξίνες σε σχέση με την απουσία αυτών των στοιχείων σε σχέση με ε, την, ε, τα ειζήματα καθώς επίσης και ε, το θέμα της υπέρβασης τιμών κατοφλίων που είναι σε χαμηλό επίπεδο. Δεδομένου αυτού του σκηνικού, αυτής της εικόνας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όταν είχαν υποβληθεί αυτά τα στοιχεία είπαμε ότι δεν υπήρχε πράγματι παραβίαση, δεν υπήρχαν επαρκή στοιχεία για να πιστούμε ότι υπήρχε παραβίαση κοινοτικής νομοθεσίας. Αυτή ήταν η δική μας θέση. Και Μόλις την προηγούμενη εβδομάδα πήραμε μια επιστολή με ημερομηνία 21 Απριλίου από τον συντάκτη. Το στείλαμε στην Επιτροπή μετά στις υπηρεσίες μετάφρασης, αλλά με μια αδρή μετάφραση σε γενικές γραμμές πιστεύω ότι αμφισβητεί ο αναφέρον τα σημεία τα οποία είχαμε εμείς αναφέρει στην τελευταία γνωστοποίηση. Υπήρχαν και κάποια στοιχεία ε, σε παράτημα, όμως εκπλήσωμε ότι έχουν ημερομηνία Δεκεμβρίου 2005. Θα ήθελα να αναφέρω ολοκληρώνοντα ότι οι υπηρεσίε τη Επιτροπή με ιδιαίτερη ικανοποίηση να εξετάσουν το θέμα αυτό επιπρόσθετα το οποίο υποβάλλει ο αναφέρον. Οι πληροφορίες που ουσιαστικά αναφέρει πράγματι θα πρέπει να εξεταστούν. Αν υπάρχουν εδώ λοιπόν κάποια στοιχεία και δεν είναι δυνατόν να υπάρξει μια ας το πω έτσι ε, συλλήβδινα απάντηση θα εξετάσουμε αυτό το θέμα και θα έρθουμε να χρειαστεί σε επαφή με τις αρμόδιες αρχές αλλά τα στοιχεία που πήραμε από τις αρμόδιες κρατικές αρχές ε, ικανοποιούν τις ε, απαιτήσεις της υπηρεσίας μας. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Άουκεν παρακαλώ. Θα ήθελα να πω ότι είναι κάπως δύσκολο για μας εξετάζοντας και βλέποντας σε ερευνητική αποστολή, για παράδειγμα αύριο το πρωί, και καθότι μπορώ εγώ να διακριβώσω από τις πληροφορίες που έχουμε από τις τοπικές αρχές ίσως μπορεί, να παρανόησα κάτι αλλά καθώς είναι ζώνη ε, παραθεριστών και ε, διακοπών είναι πολύ σημαντικό να ε, διασφαλίζεται η διάσταση αυτή για ε, την ανθρώπινη συμμετοχή σε αυτή τη ζώνη. Να μην ε, απολεστεί η προσπελασιμότητα αυτής της ζώνης, να μην αρνηθούμε πρόσβαση σε πολίτες ε, σε αυτή τη ζώνη, σε αυτή την περιοχή. Ίσως όμως μπορεί να παρανόησα την απάντησή σας. Νομίζω είναι πολύ δύσκολο να πούμε ότι όλα βαίνουν καλώς όμως θα έλεγα. Ευχαριστώ. Ναι, κατανοώ την αντίρρηση της κυρίας Άουκεν κατανοώ τις, ε, τις αντιρρήσεις σας. Είναι σαφές ότι χρειαζόμαστε περισσότερες πληροφορίες, σίγουρα. Κανονικά οι αναφερόμενοι συντάκτες αναφορών ήθιστε να υποβάλουν τέτοιου είδους στοιχεία και αναφορές. Θα χρειαζόμαστε λοιπόν τεκμηρίωση, ας το αποκαλέσω έτσι από πλευράς του αναφέροντος προτού οποιοδήποτε θα μπορούσε να αποφασίσει αν θα έπρεπε να ξεκινήσουν διαδικασίες επί παραβάση ή παραβιάση ή όχι. Εν πάση περιπτώσει, σε αυτή τη συγκεκριμένη εξειδικευμένα περίπτωση, όπως ανέφερε και ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι αναφέροντες θα μπορούσαν ίσως να μας παράσχουν περισσότερα στοιχεία ή τεκμήρια για να βασιστούμε σε αυτά σε όλα λοιπόν έχουν γίνει έσω και μέσω ανακοινέσεων ανάμεσα ε, στην Επιτροπή και στις τοπικές αρχές ε, με παρόμοιες απαντήσεις, ε, με παρόμοιες έρευνες επιβεβαιώσεις δεν μπορούμε να προχωρήσουμε περισσότερο εκτός αν έχουμε παραπάνω στοιχεία. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να προτείνω μετά από όλα αυτά που υπόθηκαν να κλείσουμε το θέμα και να ανακοινώσουμε το αποτέλεσμα των σημερινών μας εργασιών στους αναφέροντες και το τι έγινε με τις έρευνες όπως μας τα είπε η Επιτροπή. Κοιτάξτε όμως, ε, η εξήγηση που μόλις δώσατε πρέπει κάπως να την ε, καταλάβει και ο αναφέρον. Για ποιο λόγο κλείνουμε έτσι την αναφορά. Μα είπατε ότι δεν υπάρχουν ε, νέε πληροφορίε, ότι δεν έχουν προκύψει νέα στοιχεία και ότι γι' αυτό το λόγο ε, θεωρούμε ότι περατώνεται η αναφορά αυτή. Δηλαδή, αν θέλετε να το συμπεριλάβουμε αυτό στην επιστολή. Εντάξει. Τώρα έχουμε την. Μισό λεπτό να δω. Госпожо председател, извинявайте, че ще ви задам този въпрос, но искам едно малко... Кирия Проедре, κυρία Πρόεδρε, ένα ίσονος σημασία θέμα για αποσαφήνιση. Εχθές κατά τη διάρκεια της συνεδριάσεως που κάποια σημεία, 4-5 αναφορές στην ημερήσια διάταξη εχθές, δεν εξετάστηκαν τι θα κάνουμε λοιπόν, τι θα πούμε σε εκείνους τους ανθρώπους που γνωρίζουν ότι οι αναφορές τους θα εξεταζόντουσαν στην ε, δική μας Κοινοβουλευτική Επιτροπή και μετά οι, επιτρο... οι αναφορές τους αυτές καθυστέρησαν πάλι και δεν εξετάστηκαν και πάλι. Κάποιες εκκρεμούσαν τα τελευταία τρία χρόνια για να εξεταστούν. Τι θα πούμε και πώς θα ισχυριστούμε ότι, είμαστε, ότι υπάρχει αξιοπιστία σε σχέση με τους πολίτες μας και εμπιστοσύνη όταν ακολουθούμε τέτοιου είδους διαδικασία. Ε, e- Εντάξει, το δέχομαι, το επιβεβαιώνω, να το διορθώσω ίσως όχι από το 21, δεν θα έπρεπε από εκεί να αρχίσουμε, αλλά από εκείνα που είχαμε αναβάλει για να έχουμε πρώτα τις αναφόρες ε, που είχαμε και παρόντες τους αναφέροντες. Εάν σήμερα δεν τα καταφέρουμε να εξετάσουμε αυτές τις αναφορές που αναβάλαμε, τότε θα στείλουμε γραπτή απάντηση στους αναφέροντες, θα το κάνουμε την επόμενη φορά και θα πάνε για την επόμενη συνεδρίασή μας αυτές. Θα προσπαθήσουμε όμως, σας διαβεβαιώνω, να τις εξετάσουμε ήδη σήμερα. Επιτρέψτε μου να διαφωνήσω, Πρόεδρε. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Επειδή Πολλοί από αυτούς με τους οποίους ήρθα σε επαφή χθε κιόλα, τους αναφέροντες δεν είχαν ενημερωθεί από τη γραμματεία μας ότι η αναφορά τους είχε εγγραφεί στη χθεσινή συνεδρίαση και δεν είχαν προσκληθεί καν να είναι παρόντες. Αυτό είναι πραγματικά συγχώρητη έλλειψη και θα πρέπει να υπάρξουν συνέπειες νομίζω να μην γίνει κάτι τέτοιο. Για πρώτη φορά μου γνωστοποιείται αυτό. Εάν οι αναφέροντες, όπως μας λέτε, δεν ειδοποιήθηκαν, τότε ακόμα περισσότερο ισχύει το ότι δεν θα πρέπει να εξεταστούν οι αναφορές αυτές τώρα. Να τους ενημερώσουμε και ενδεχόμενα να τους καλέσουμε να συμμετάσχουν στις εργασίες της Επιτροπής και μετά να αναβάλουμε την εξέταση για την επόμενη φορά. Μήπως η Γραμματεία κάτι θα ήθελε να προσθέσει σχετικά, γιατί δεν ενημερώθηκαν οι αναφέροντες τι συνέβη. Uh, θα προσπαθήσουμε προφανώς και θα έρθουμε σε επαφή με τους αναφέροντες. Ζητούμε συγγνώμη για το ότι δεν έγινε αυτό όταν θα διασφαλίσουμε ότι θα εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη όσο το δυνατόν νωρίτερα αν γίνεται. Σα Σας ευχαριστώ. Εμένω και επιμένω όμως αυτό να μπορέσει να γίνει αμέσως στην επόμενη συνεδρίασή μας. Θέματα τεράστια σημασία είναι αυτά. Όλη τη μέρα χθε την αναλώσαμε συζητώντας ειδικέ ανάγκες για, άτομα και θα είναι ασυγχώρητη έλλειψη αν αυτό δεν καλυφθεί και δεν μπορέσει να εξεταστεί την επόμενη συνεδρίασή μας. Ε, Καλό και σωστό θα ήταν να γίνει την επόμενη συνάντηση. Θα είμαστε όμως σε θέση να το κάνουμε αυτό τότε. Γιατί έχουμε καλέσει και την ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή τις επόμενες, την επόμενη φορά πολλά μπήκαν το ένα μαζί με άλλο. Έχουμε πολύ λίγο χρονικό διάστημα στη διάθεσή μας ε, για να έχουμε την παρουσία αυτής της Επιτροπής, να έχουμε τους ε, αναφέροντες κλπ. Τέλος πάντων, την επόμενη εβδομάδα θα προτείνω εγώ στην ομάδα των συντονιστών τι μπορεί να γίνει για να αλλάξουμε αν γίνεται την ημερήσια διάταξη της επόμενης συνάντησης της Επιτροπής 31 ε, Μαΐου, 1 Ιουνίου και έτσι να μπορέσουν να συμμετάσχουν οι αναφέροντες αν γίνεται, αν γίνεται την επόμενη φορά, την επόμενη μας συνάντηση. Eh, Αυτά. Να προχωρήσω λοιπόν. Έχουμε όλες τις εκθέσεις που αναβάλαμε χθες. Για να δούμε. Συνάδελφε, Πέστε μου sworn Yes, but we can change. We can change it. We have the power to change it. We can have a look at it, but it needs to be. It was the coordinators that decided. Λοιπόν, συγγνώμη για τη διακοπή. Να ξεκινήσουμε και πάλι αυτή τη φορά από το σημείο 29. Έχει δοθεί ο λόγο από πλευρά συναδελφού Βίλαντ. Ήθελε να αλλάξει με το 28 για να είναι. Για, να υπάρχει παρουσία. λοιπόν, πάμε στην 29. Νάιντεν Σαχάροφ, βουλερική Ιθαγένεια. Η Επιτροπή. Σα ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αυτή η αναφορά αφορά τους όρους λειτουργίας μιας μονάδας ε, παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ε, στην Μαρίτσα η στη Βουλγαρία. Γνωρίζει πολύ καλά αυτή την εγκατάσταση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την αξιολόγηση για την αδειοδότηση που έγινε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Με βάση αυτήν την αξιολόγηση βρέθηκε ότι η άδεια ευθυγραμμίζεται με τις απαιτήσει της IPPC για την πρόληψη και καταπολέμηση της μόλυσης καθώς επίσης και για τους όρους καύσης. Οι όροι για την λειτουργία αυτή και την άδεια εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των αρμόδιων αρχών στο κράτος μέλος. Ίσως θα μπορούσε πράγματι να είναι διαφορετική η πραγματικότητα από αυτή που αναφέρεται και εμπεριέχεται στην άδεια λειτουργίας. Αλλά αυτό θα πρέπει είναι θέμα θέμα του αρμόδιου κράτους. Επιπλέον, ε, όσον αφορά τον μη σεβασμό των ε, ε, κατοφλίων τιμών όσον αφορά τη μόλυση του περιβάλλοντος, μια διαδικασία παραβάση παραβάσει έχει ξεκινήσει. Είναι γνωστό ότι οι τιμές αυτές της Βασιλείας 2 δεν γίνονται σεβαστές σε σχέση με αυτές τις ζώνες και για τη Μαρίτσα Ίστοκ και τη ζώνη αυτή λαμβάνεται δράση, αναλαμβάνεται δράση λοιπόν κατά της Βουλγαρίας ε, λόγω αυτής της παράβασης. Ευχαριστώ. Κοιτάξτε, νομίζω ότι πρέπει να το αναβάλουμε μέχρι να λάβουμε την απάντηση τα αποτελέσματα. Εντάξει, αφήνουμε ανοιχτό το θέμα για να δούμε τι γίνεται με αυτή τη διαδικασία που έχει ξεκινήσει. Το επόμενο είναι το 30 1501 2008 της Διονυσίας Αυγερινοπούλου ελληνική Ιθαγένειας. Φλόιντ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε η ε, ε, αναφέρουσα έχει υποβάλει και ε, προσφυγή και όσον αφορά τις εξοριστικές δραστηριότητες στην Μήλο και καθώς θα δείτε από προηγούμενη πληροφόρηση πολλές από τις, πολλοί από τους ισχυρισμού σε σχέση με αυτή την προσφυγή δεν μπόρεσαν να τύχουν συνέχεια με εξαίρεση ένα θέμα την δυνατότητα της φόρτωσης επικίνδυνων ουσιών στο υδάτινο περιβάλλον. Ε, θίξαμε το θέμα αυτό στις ελληνικές αρχές που επίσημα πίντησαν και ακόμα και όταν έχουμε περλίτη και μπεντονίτη που εξορίσσονται είναι ε, πιθανό να υπάρχει και ε, περιεκτικότητα σε νικέλιο και σε ανάλυση των υδάτων η ανάλυση το, το αποτέλεσμα ήταν ότι ήταν καλύτερο και από την ποιότητα του πόσιμου ύδατος. Λοιπόν, αυτό σε σχέση με, αυτή την, με, αυτό το επιχείρημα. Είπε η αναφέρουσα ότι θα επανερχόταν σε σχέση με το θέμα αυτό σε επαφή μαζί μας. Δεν το έκανε. Ίσως σε σχέση ακριβώς με αυτό θα ε, ήταν σκόπιμο να κλείσει η αναφορά. Παρότι μας είπε ότι θα υπέβαλε νέα στοιχεία σε ανακοίνωση που θα υπέβαλε, δεν το έκανε η αναφέρουσα. Συμβαίνει καμιά φορά συντάκτες αναφορών ή ε, ε, προσφεύγοντες ε, να καταλήγουν σε αυτό. Αυτό είναι το οποίο συνέβη τώρα εδώ. Ευχαριστώ. Ehm, η πρόθεση αυτή δεν φαίνεται καθαρά, δεν ξέρω για περαιτέρω στοιχεία. Βλέπω όμως και στην απάντηση ότι από την Επιτροπή δεν υπήρξε σαφήνεια. Τέλος πάντων, σας λέω συνάδελφοι ότι η συνάδελφος κύριε Παλιαδέλη είχε ζητήσει να παραμείνει ανοιχτή αυτή η αναφορά γιατί χρειαζόταν και περαιτέρω στοιχεία. Άρα λοιπόν αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις παραμένει ανοιχτό το θέμα επειδή το έχει και επειδή δεν έχει δώσει εξαντλητική απάντηση η Επιτροπή. Συμφωνώ απολύτως ε, και θα ήθελα να προσθέσω ε, ότι έχουμε ούτως ή άλλως ε, υπόψη μας να εξετάσουμε αυτό το θέμα της επεξεργασίας αποβλήτων στην Ελλάδα. Είναι ένα παλιό θέμα και νομίζω ότι είναι πολύ καλό να διατηρήσουμε εκρεμή την αναφορά αυτή. 31 τώρα. Τζόνα Μολίνσκα, Πολωνική ηθαγένεια. Ο εκπρόσωπο τη Ευρωπαϊκής Επιτροπή Φρανσουά Κρέμα, έχει το λόγο. Ε, Ευχαριστώ πολύ. Πρόκειται για την ε, εκμετάλλευση ενός ε, λατομείου στην Πολωνία. Δεν θα σας πω το όνομα γιατί είναι λίγο περίπλοκο. Ήρθαμε σε επαφή με τις πολωνικές αρχές για το θέμα αυτό και η απάντηση που λάβαμε είναι ότι οι δραστηριότητες του λατομείου έχουν διακοπή κυρίως γιατί ούτως ή άλλως το πρόγραμμα των δραστηριοτήτων ε, δεν ήταν συμβατό με το πρόγραμμα χωροταξίας της περιοχής ε, και υπάρχουν δύο πτυχές αυτήν την αναφορά. Πρώτον, ε, οι δραστηριότητες εκμετάλλευσης του λατομείου που έχουν ήδη ξεκινήσει και επίσης ένα πρόγραμμα επέκτασης των δραστηριοτήτων του λατομείου αυτού. Αυτά τα δύο ζητήματα διέπονται βέβαια από την εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων και διέπονται και από την οδηγία ε, για το οικοσύστημα και την, το Natura 2000. Το γεγονός ότι διεκόπησαν οι ε, δραστηριότητες ε, είναι μια επιτυχία. Επιμείναμε στις πολωνικές αρχές ε, και ειδικότερα για το σεβασμό των διατάξεων των δύο οδηγιών σε σχέση με την ε, επέκταση ε, του λατομείου και ενημερώσαμε επίσης ε, μία ακόμη φορά για την ανάγκη σεβασμού των ε, διατάξεων και θα το ξανοκάνουμε όταν επαναλάβει τις δραστηριότητες το εν λόγω λατομείο θα επιβεβαιώσουμε κατά πόσο έχουν γίνει σεβαστές ε, οι διατάξεις αυτές και αν όχι θα ξεκινήσουμε διαδικασία επιπαραβάση. Μπορούμε να αφήσουμε κρεμή πιστεύω την αναφορά αυτή μέχρι να υπάρξουν περαιτέρω εξελίξεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Όκεν. Αυτή τη φορά νομίζω ότι πρέπει πραγματικά να επενέσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Με μεγάλη χαρά θα το κάνω. Να τους επενέσω, να τους πω ότι ήταν καταπληκτικοί. Να μας ενημερώσετε, να μας ενημερώσετε. Ευχαριστούμε. Καταλαβαίνω λοιπόν ότι θα αφήσουμε ανοιχτό το θέμα και θα παρακολουθήσουμε με ιδιαίτερη προσοχή την εργασία της Επιτροπής. Ε, τελευταία η 32, 884, 2009 Βρετανικής Ιθαγένειας ο αναφέρον, ο εκπρόσωπο τη Επιτροπής. Μπλόχ. Ευχαριστώ. Αυτή η αναφορά αφορά ένα παράπονο πολίτη από την Ουαλία σε σχέση με την ε, χρήση ε, του αποχετευτικού δικτύου και την ε, δυσοσμία και τους κινδύνους που απορρέουν για τους περίκους. Γραπτός υπήρξε ενημέρωση σε σχέση με τις νομικές διατάξεις που επιβάλλονται από το δίκαιο στο Ηνωμένο Βασίλειο. Τα καλά μαντάτα όμως φαίνεται ότι είναι λίγες μέρες πριν από την παράληψη αυτής της προτού λάβει αυτή την αναφορά η Επιτροπή, οι τοπικές αρχές στο τοπικό συμβούλιο κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι τα αναγκαία διαβήματα είχαν ήδη γίνει από την ε, τοπική υπηρεσία υδάτων και υπέβαλε έτοιμα ε, να την συγχωρέσουν οι πολίτες ε, για τα προβλήματα τα οποία έπρεπε να υποστούν επί κάποιο χρονικό διάστημα. Από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα αναγκαία μέτρα έχουν ήδη ληφθεί. Πρέπει όμω να πούμε με κάποια καθυστέρηση, διότι υπήρχαν παράπονα των πολιτών ήδη το 2003 και το 2004 για αυτή την κατάσταση. Αυτή τη στιγμή φαίνεται λοιπόν ότι τα αναγκαία βήματα έχουν γίνει και δεν προβλέπει ανάληψη περαιτέρω δράσεως σε αυτή τη χρονική συγκυρία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Λοιπόν, κλείνει το θέμα της αναφοράς αυτής. Θεωρούμε ικανοποιητική την, αποφα... την απάντηση της Επιτροπής. Τελευταία, 28, πως Βίλαντ είχε ζητήσει ακριβώς να καθυστερήσουμε, παρ' αυτά δεν παρίσταται. Λοιπόν, η 181-2009 Καρλ ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε σε αυτήν εδώ την αναφορά που είναι μια αναφορά που ήδη στη Βάδη Βιρτεμβέργη στο Κοινοβούλιο είχε υποβληθεί στο, στην τοπική βουλή επρόκειτο για την εξέταση θεωρούμε εμείς κατά πόσον εδώ έχει παραβιαστεί το κοινοτικό δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, περί τίνος πρόκειται εδώ. Ο αναφέρον παραπονείται ότι στη δική του περιοχή, στη δική του γειτονιά δημιουργήθηκε μια μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που με βάση τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας εδώ ήταν το φινικέλαιο ως πρώτη ύλη όπου αρχικά είχε βέβαια προβλεφθεί εδώ να μπορούν να λειτουργήσουν και συσκευές που όμως από πλευράς διεργασίας μειώθηκαν σε μία τέτοια συσκευή και στη συνέχεια ε, ακολούθησε η πρόσθεση δεύτερης εδώ δεν έγιναν μελέτες περιβαλλοντικής συμβατότητας για λόγους που όσον αφορά τις τιμές κατόφλια που σύμφωνα με το γερμανικό δίκαιο θα έπρεπε να είναι σεβαστές δεν μπόρεσαν να επιτευχθούν. Δηλαδή η μονάδα και, το, και επιπλέον αυτή η συσκευή ήταν κάτω από ένα μεγαβάτ ε, παραγωγής ε, ενέργειας, απόδοσης ενεργειακής. Γι' αυτό δεν μπορούσαμε εδώ να διαπιστώσουμε παραβίαση ε, νομικών διατάξεων του ευρωπαϊκού δικαίου διότι σε σχέση με τα κράτη-μέλη όσον αφορά την ε, οδηγία συμβατότητας ε, προβλέπεται η ευθυγράμμιση και συμμόρφωση σε σχέση με τα στοιχεία στο παράρτημα 1 και εδώ δεν είναι υποχρεωτική μια τέτοια μελέτη συμβατότητας είτε για τον καθορισμό κατώτατων τιμών είτε για την αναπερίπτωση εξε, εξέταση ή και με συνδυασμό των δύο διαδικασιών να μπορέσει να διαπιστωθεί αν θα πρέπει να γίνει μια τέτοια εξέταση ή όχι. Σύμφωνα με το παράτημα 1 θα ήταν σαν συνέπεια τούτου ε, ε αναγκαίο να εξετάσουν οι αρμόδιες αρχές ε, αν αυτές οι εγκαταστάσεις ε, και τα στοιχεία τους θα ήταν τόσο σημαντικά ώστε να απαιτείται μια πλήρης αξιολόγηση ή όχι. Αυτή η προεξέταση δεν έγινε, διότι σύμφωνα με το γερμανικό δίκαιο αυτή η μονάδα παραμένει κάτω από την επίδοση ενός ΜΒ. Όμως το κυριότερο στοιχείο αυτής της αναφοράς είναι ότι ο αναφέρον θεωρεί ότι πρόκειται για μια συνδεδεμένη μονάδα, διότι εδώ δύο γεννήτριες εργάζονται συνδεδεμένες από κοινού. Μόνο που τώρα ο κάθε, η κάθε γεννήτρια σύμφωνα με τον αναφέροντα είναι αντικείμενο εκμετάλλευσης από μια ΕΠΕ, μια εταιρεία ε, εταιρεία περιορισμένης ευθύνης και λέει ότι εδώ πρόκειται για μια ας πω έτσι υπόθεση που κάθε εταιρεία έχει έναν, μια γεννήτρια που εκμεταλλεύεται. Πρέπει όμως από κοινού να εξετάζονται αυτές οι δύο γεννήτριες και έτσι συνδεδεμένες όταν λειτουργούν ξεπερνούν, ε, θα φτάνανε στο 1 ΜΒ και θα έπρεπε να ε, ακολουθήσει η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Όλα αυτά όμως είναι θέματα αποκλειστικά εφαρμογή εφαρμογής εθνικού δικαίου και όχι ευρωπαϊκού δικαίου. Για αυτή τη μονάδα σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες υπάρχει μια άδεια λειτουργίας, μια άδεια λειτουργίας που όπως είναι φυσικό θα πρέπει να, είναι, να καθορίζει ότι οι εκπομπές ρήπων αυτών, αυτής της μονάδας θα ανταποκρίνονται απόλυτα με τις ε, προδιαγραφές του ενισχύ δικαίου. Από ό,τι γνωρίζουμε ο αναφέρον υπέβαλε προσφυγή στο διοικητικό δικαστήριο για αυτή την απόφαση ωστόσο όμως το διοικητικό δικαστήριο δεν έκανε δεκτή την προσφυγή του την κατηγορία αυτή. Εμείς ως συμπέρασμα αναφέραμε αν είναι σε θέση ο αναφέρον να υποβάλει περαιτέρω στοιχεία σε εμά για τους λόγους που θα μπορούσαν να είναι πιστικότεροι και θα μπορούσαν να δείξουν ότι υπάρχει λόγος ανησυχίας για την, ε, ε, ε, όσον αφορά μέσα ρήπων και όσον αφορά το ευρωπαϊκό δίκαιο, όσον αφορά τις εκπομπές ρήπων, αυτό θα το ξαναβλέπαμε, είπαμε. Αν όμως ε, σύμφωνα με το, την υποβολή στοιχείων καταδεικνύεται ότι πρόκειται για την προσπάθεια για την παράκαμψη μιας ε, ας αποφυγή όρων που πρέπει να σέβεται μια τέτοια ε, μονάδα. Αν εδώ πρόκειται δηλαδή για μια προσπάθεια να ε, παρακαμφθεί κάποια διάταξη θα έπρεπε να δώσουμε συνέχεια. Όμως εδώ και σύμφωνα με το ε, γερμανικό δίκαιο ε, δεν θα έπρεπε από τις αρμόδιες αρχές με, μετά από προσφυγή να ισχύσει το εθνικό δίκαιο και πάλι και οι διατάξεις του όσον αφορά αυτό το θέμα. Συνοψίζω, αν ο αναφέρον μας δώσει νέα, μας έδινε νέα στοιχεία ή πιο εξειδικευμένα, τεκμηριωμένα στοιχεία ότι αναφέρεται σε σχέση με την αναφορά του σε θέμα που αφορά το ευρωπαϊκό δίκαιο, τότε θα εξετάζαμε το θέμα αυτό σε μεγαλύτερο βάθος. Δεν μπορούμε όμως να ασκήσουμε επικρίσεις όταν τα κράτη-μέλη ασκούν τα δικαιώματά τους όσον αφορά τέτοια θέματα και τιμές κατοφλίου εκπομπών ρήπων σε σχέση με το όπως έχουν σήμερα τα πράγματα θα έπρεπε με την λειτουργία δύο ξεχωριστών συσκευών όπως έχει προβλεφθεί εδώ να διαπιστωθεί ότι υπάρχουν συσσωρευτικές τέτοιες επιπτώσεις στο περιβάλλον. Και σε περίπτωση που θα συνέβαινε κάτι τέτοιο θα έπρεπε να γίνει μια προεξέταση από πλευρά των αρχών. Αυτό όμως απομένει να αποδειχθεί. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε γνώριζα ότι θα ήθελε να έρθει ο αναφέρον εδώ και θα είχαμε μια ευκαιρία να το συζητούσαμε. Αλλά εντάξει, ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Γιάρ, παρακαλώ θα ήθελα το συμπέρασμα να το συμπληρώσω σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όχι μόνο να δύο αναφέρον αν μπορεί περαιτέρω στοιχεία και τεκμήρια να προσθέσει για την αναφορά του, αλλά και να αποστείλει επιστολή στην αρμόδια αρχή στην ε, ε, Γερμανία. Κάπως ακατανόητα μου φαινόντουσαν αυτά τα οποία είχαν συνταχθεί διότι είχαμε τεράστια αντιπαράθεση στην Γερμανία για το βιοαέριο αέριο όταν πρόκειται για τέτοιες μικρές ε, τώρα εγκαταστάσεις ε, και που ε, υποστηρίζονται υπάρχουν κάποιοι εκμεταλλευτές τέτοιων ε, μονάδων που κατακαιρματίζουν τις μονάδες αυτές σε επιμέρους τμήματα. Ε, όμως ως σύνολο θα πρέπει να εξετάζονται αυτές ε, οι μονάδες. Πρόκειται λοιπόν εδώ και να το γνωρίζουμε αυτό για ένα τέτοιο σύνολο εγώ δεν μπορώ να το τεκμηριώσω αυτό. Ίσως θα πρέπει οι αρχές ε, πρώτα να τοποθετηθούν ε, πώς καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για δύο ξεχωριστές μονάδες ε, ή κατά πόσον αυτές συνδέονται ή όχι. Εγώ δεν μπορώ να το κρίνω αυτό από αυτή την αναφορά. Και όχι μόνο σε σχέση με τον αναφέροντα, αλλά και η τοπική αρχή, η κρατική αρχή θα έπρεπε να τοποθετηθεί από αυτού. Ίσως υπάρχει το αποτέλεσμα εντωμεταξύ σε σχέση με την Επιτροπή Αναφορών του Κρατηδίου της Βάδης Βιρτεμβέργης γι' αυτό. Σε σχέση με την παρουσίαση θα έλεγα όλα είναι κάπως αξιοπε... αξιοπερίεργα και αλόκοτα θα έλεγα. Ευχαριστώ. Ναι, έχει δοθεί οτιδήποτε με, το, με, διάφορα στοιχεία. Έτσι μπορεί να δείτε τι ακριβώς γίνεται. Απλώ ήθελα να πω ότι συμφωνώ με τον Πίτερ Γιάρ και εμένα μου έκανε λίγο εντύπωση από την αρχή όταν άκουσα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μόνο αν υπήρχε πρόθεση διάσπασης της μονάδας, δηλαδή θα μας, θα μας απασχολούσε, θα μας ενδιέφερε το θέμα αλλά θα μας ενδιέφερε μόνο, θα μας ενδιέφερε και ακόμη και αν ε, ε, ήταν ε, τυχαίο. Ακόμη και αν δεν υπήρχε πρόθεση δηλαδή διέρεσης, από τη διαίρεση της μονάδας παραγωγής. Ας περιμένουμε λοιπόν περαιτέρω στοιχεία. Παραμένει ανοιχτό το θέμα αυτό για αυτή την αναφορά και έτσι ανταποκρινόμαστε σε αυτό που είπε ο συνάδελφος για να μπορούμε να συμμετάσχουμε και να βοηθήσουμε. Ολοκληρώσαμε έτσι τις εργασίες μας. Θα σας ευχαριστήσω. Γεια σας. Θα τα πούμε την επόμενη συνεδρίασή μας.